Παρακαλώ τους συναδέλφους από τις μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες να καλέσουν τους συναδέλφους, κυρίως συντονιστές, για να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Έχουμε, έχουν ήδη παρέλθει 10 λεπτά. Είναι νομίζω λογική καθυστέρηση. Ε, πάνω από 10 λεπτά όμως δεν θα ήταν λογική καθυστέρηση. Προχωρώ λοιπόν. Και ξεκινάμε τη συνεδρίασή μας. Σε κρυσιμερησία διατάξεις υπάρχουν προτάσεις, αντιρρήσεις. Ε, εγκρίνεται πρακτικά της ε, τελευταίας μας συνεδρίασης 29 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου ως ήθιστε θεωρούνται πως εγκρίθηκαν εάν δεν υπάρχουν έως το τέλος της ε, συνεδρίας ως Στο σημείο 3 συνήθεις ανακοινώσεις, ότι έχουμε δηλαδή μετάδοση από το διαδίκτυο της ε, συνεδρίασής μας και κατάλογος ε, αλληλογραφίας για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται. Πριν περάσουμε στην ουσία όμως της συνεδριάσεως μας, θα ήθελα να συγχαρώ το Γιάρος Λεβαρένσα, το φίλο μας που ξανάρθε. Και πάλι καλά, γερός και δυνατός μετά το ατύχημά του. Μας έλειψες. Καλώς ήρθες. Και έχουμε και ένα νέο συνάδελφο, τον κύριο Αμιά Αμπάντα. Από την Επιτροπή των Προϋπολογισμών, εάν δεν απατώμε. Και ήταν πολύ σοφή η απόφαση να έρθεις σε μας. Νομίζω ότι θα βρεις πολύ ενδιαφέρουσα στις συνεδριάσεις μας. Ας περάσουμε τώρα στην ουσία της σου, στο σημείο 5. Αντικείμενα δι, διπλής χρήσης. Όχι. Είναι το σημείο 4 καταρχάς. Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων της Επιτροπής μας. Παρακαλώ. Αυτό είναι μια επιλογή η οποία σε στόχο έχει να ε, αξιοποιούμε πιο λογικά, πιο ορθολογικά τις υπηρεσίες διερμηνίας για να έχουμε λιγότερη ε, σύμπτωση συνεδριάσεων σε μία-δύο μέρες μόνο. Άρα, οι συνεδριάσεις επιτροπής μας θα πρέπει να γίνονται ή Δευτέρα απόγευμα με Τρίτη απόγευμα, τρεις μισές μέρες δηλαδή, ή από Τετάρτη πρωί μέχρι Πέμπτη απόγευμα. Επαναλαμβάνω. Πέμπτη απόγευμα. Εάν θέλουμε να έχουμε τέσσερις μισές ημέρες, δύο πλήρες ημέρες συνεδρίες. Και όλα αυτά είναι σοβαρές υποθέσεις. Έχουμε το νέο χρονοδιάγραμμα λοιπόν, με μόνη αλλαγή που αναγκαστικά εισάγεται είναι στην εβδομάδα υπαριθμών 38 η έναρξη συνεδριάσεως τη Δευτέρα το απόγευμα. Άρα, προς το παρόν, πέμπτη απόγευμα δεν έχουμε. Πλήνω. Μια ιδέα που θα σας προτείνω αργότερα. Στο σημείο 5, λοιπόν, ήδη διπλής χρήσης. Όπως γνωρίζετε, πρόκειται για ένα θέμα το οποίο για δεύτερη φορά μας απασχολεί. Πρόκειται για εξέταση ενός κανονισμού του Συμβουλίου και σε δεύτερη ανάγνωση. Όπως ξέρετε έχω εγώ αναλάβει και ως εκ τούτου θα σας παρουσιάσω αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις το θέμα αυτό ως εισηγητής πλέον. Δεν βλέπω αντιρρήσεις. Όπως ορίζετε λοιπόν η Επιτροπή μας Φαντάζομαι ότι έχετε δει στον φάκελο τα, κείμενα, δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε, έχει αποφασίσει να αξιοποιήσει την υφιστάμενη νομοθετική διαδικασία η Επιτροπή μας για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη διαδικασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα είδη διπλής χρήσης, ύστερα από την απόφαση πέρσι ε, ε, τη σχετική με τα συστήματα ελέγχων. Προτείνω λοιπόν την έγκριση των θέσεων, της θέσεως του Συμβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση από το Συμβούλιο, από το Κοινοβούλιο. Αυτή είναι η πρότασή μου. Είναι ένα τεχνικό θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να δεχθεί το χαρακτηρισμό διπλής χρήσης των εξωτερικών διεθνών οργάνων, κυρίως σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών. Και άρα έτσι επικαιροποιείται ο κατάλογος ο δικός μας, ο νομοθετικός κατάλογος και προσαρμοζόμαστε στις επιλογές των παγκοσμίων φορέων. Άρα διακριτική ευχαίρεια δεν υπάρχει εδώ, πλην της ευθυγράμμισης της νομοθεσίας μας με τις αποφάσεις των διεθνών φορέων στον τομέα αυτό και αυτό είναι το ε, κείμενο, αυτή είναι η πρότασή μου. Προτείνω λοιπόν να θετήθει η θέση του Συμβουλίου σε... από την πρώτη ανάγνωση. Και αυτό είναι όλο. Είναι ο πιο ταχύς τρόπος λοιπόν να προχωρήσουμε. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις. αντιρρήσεις, σχόλια. Χρόνο διάγραμμα. Θα ψηφίσουμε εδώ αύριο και 29 Μαρτίου στην Ολομέλεια. Άρα παρακαλώ να είστε ενήμεροι να θυμάστε ότι αύριο ψηφίσουμε το θέμα αυτό στην Επιτροπή μας. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, το υπαριθμόν 6. Ο κύριος Βίγκλερ από το ΕΛΚ με παρακάλεσε να τον αντικαταστήσει ο κύριος Γκάσπαρη, γιατί ο κύριος Βίγκλερ δεν μπορούσε να έρθει, αλλά λείπει και ο κύριος Γκάσπαρη, οπότε προχωρούμε πιο πέρα, μέχρι να έρθει ο κύριος Γκάσπαρη, και οπότε θα, και θα επιστρέψουμε στο σημείο 6. Στο 7 μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή σε τρίτες χώρες. Καταρχάς έχουμε την παρουσίαση μιας μελέτης και δεύτερον έχουμε εξέταση ενός σχεδίου εκθέσεως. Είμαστε αρμόδια ουσία επιτροπή με εισηγητή τον κύριο Καζάκ. Θα πρότεινα λοιπόν να δούμε την κριτική εκτίμηση εδώ, την μελέτη που σας δείχνω σε έντυπη μορφή που έχετε στη διάθεσή σας, όπως και το κοινό γενικότερα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μάικλ Έμερσον, που είναι Όχι. Μάλιστα. Δεν είναι εδώ, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε την παρουσίαση της μελέτης. Τι να κάνουμε τώρα, να αφήσουμε και την εξή του σχεδίου εκθέσεως από τον εισηγητή μας. Να δούμε την παρουσίαση. Με τι είναι άλλο. Επομένως, αντί για δεύτερο τμήμα, έρχεσαι τώρα εσύ να κάνεις την παρουσίαση της μελέτης σου, της, ε, την εξέταση του σχεδίου με έκθεσης. Έχετε το κείμενο της εκθέσεως. Πολλές σελίδες, το συγγνώμη για τον πέρδεμα. Ας ακούσουμε λοιπόν τον εισηγητή. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καλωσορίζω την ευκαιρία της συζήτησης, τη συζήτηση του σχεδίου εκθέσεως και ενδεχομένως της μελέτης για τον κανονισμό πλαίσιο για μακροοικονομική ενίσχυση. Θα είδατε το έγγραφο εργασία. Το σχέδιο εκθέσεως επίσης. Άρα δεν θα αναφερθώ στις λεπτομέρειές τους, όμως θα ήθελα να αναφέρω κάποια πράγματα, βασικές ιδέες. Πρώτα απ' όλα, κάποια κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με την έκθεση. Η χρήση των κατουξιδότησιν πράξεων. Πρώτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι κατά περίπτωση οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται μέσω εφαρμοστικών πράξεων για να επιταχυνθεί η διαδικασία λήψης ε, αποφάσεων. Όπως προανέφερα στην Επιτροπή, η χρήση εφαρμοστικών πράξεων δεν είναι αποδεκτή. Και αυτή είναι η κόκκινη γραμμή για μένα που είμαι ο εισηγητή. Όμω καταλαβαίνω τι ανησυχίε που εκφράζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την αποδοτικότητα ε, τη ε, οικονομική αυτή βοήθεια που υποτίθεται ότι είναι ένα μέτρο έκτακτη ανάγκη. Εξέφρασα προθυμία, όπως και η Γραμματεία, να συνεργαστούμε με τη νομική υπηρεσία για να δούμε πώς μπορούμε να χειριστούμε το θέμα. Έχω εισαγάγει το παράρτημα 2α που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τις εξουσιοδότητες συμπράξεις κατά περίπτωση όσον αφορά τις συμφωνίες. Έτσι, κατά την άποψή μου, μπορεί να ασκεί αποτελεσματικό δημοκρατικό έλεγχο το Κοινοβούλιο και το μέσο γίνεται ταχύτερο και αποτελεσματικότερο που είναι επιθυμία πολλών ενδιαφερομένων. Από την πολιτική σκοπιά. Και οι DG και οι μελέτες το, της DG Expo και η δική μου άποψη είναι ότι πολύ συχνά χορηγείται αυτή η μικροοικονομική ενίσχυση χωρίς να μην χρησιμοποιούνται τα κριτήρια του ζεμβάλου όπως αποκαλούνται. Δηλαδή ότι οι αποδέκτες της βοήθειας θα πρέπει να σέβονται ε, δημοκρατικούς μηχανισμούς. Αυτή η μικροοικονομική βοήθεια θα πρέπει να ακολουθεί τι αρχέ τη συνθήκη τη Αβώνα. Πρέπει να υπάρχει συνοχή των πολιτικών μεταξύ των συμφωνιών και των στόχων τη εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ για την πρόθεση των δημοκρατικών αρχών. Και πρέπει να προσπιστούμε τα δημοκρατικά συμφέροντα και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, στο άρθρο 6, ε, αναφέρεται ότι έχει μεγάλη δύναμη, στο σημείο 1, και ότι Πρέπει κάθε χώρα να εφαρμόζει σωστά τους δημοκρατικούς μηχανισμούς, κάθε επιλέξιμη χώρα. Μόνο αν η υπηρεσία η Ευρωπαϊκή Εξωτερικής Δράσης τοποθετηθεί θετικά θα πρέπει να επικυρώνεται η συμφωνία, να εγκρίνεται η συμφωνία. Στο άρθρο 6.4α έχω εισαγάγει μια άλλη δυνατότητα. Τα μέτρα πολιτικής και δημοκρατικής πολιτικής σύμφωνα με το Μνημόνιο ε, Συνεννόησης να εφαρμόζονται. Την περασμένη εβδομάδα πήγα στην συνεδρία τη Επιτροπή ΑΦΕΤ και υπήρχε μια πρόταση εκεί. Μια αγνομοδότηση τη Επιτροπή αυτή που ακολουθεί παρόμοιε γραμμέ. Να συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και να είναι πιο σημαντική συμμετοχή της στη λήψη αποφάσεων. Όσον αφορά το πεδίο που καλύπτεται τον κανονισμό και ποιες χώρες καλύπτει, πρώτη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρχει τρίτη κατηγορία χωρών που δεν είναι ούτε υποψήφιες ούτε χώρες γειτονίας αλλά πολιτικός, οικονομικός και γεωγραφικός είναι πλησίον της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Στην πράξη αφορά τις δημοκρατίες Κεντρικής Ασίας. Και θα πρέπει να προσθέσουμε, πιστεύω, αυτές τις δημοκρατίες σαν μια τρίτη κατηγορία. Καλύτερο αυτό παρά να έχουμε ένα όριστο και ανοιχτό ε, σύστημα για την μικροοικονομική αυτή ενίσχυση. Πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι προσωρινός αυτός ο κανονισμός με διάρκεια μόνο αυτό το οικονομικό πλαίσιο. Όμως, αυτό θα θεωρεί το παράδοξο και θα σήμαινε ότι ο κανονισμός θα ετίθεται σε ισχύ ε, για λιγότερο από δύο χρόνια. Γι' αυτό πρότεινα ο κανονισμός να μην έχει μερομηνία λήξης. Με ρήτρα αναθεώρησης βεβαίως, και έτσι θα υπάρχει νομική συνέπεια και συνοχή στον τον κανονισμό και θα αποφύγεται τυχόν αλληλεπικάλυψη εργασιών. Τέλος, για τις εκκρεμούσες διαπραγματεύσεις με τη Γεωργία για μικροοικονομική ενίσχυση, συμφωνώ με τον εισηγητή, τον κύριο Παρέδα, τον πρόεδρο, να χρησιμοποιηθεί η συμβουλευτική διαδικασία για το μνημόνιο συνεννόησης και ελπίζω να βρεθεί μια λύση που να ικανοποιεί το Κοινοβούλιο και αυτό να συμβεί στο εγγύς μέλλον. Και εδώ ολοκληρώνω την παρουσίασή μου και τα σχόλιά μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την παρουσίαση του σχεδίου εκθέσεως, λέει ο Πρόεδρος. Τα άλλα μέλη της Επιτροπής. Η κυρία Κοπά από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είχα τονίσει και στην προηγούμενη συζήτηση... Okay. You should. <laughs> It's okay. Όπως είχα τονίσει και στην προηγούμενη συζήτηση, συμφωνώ, απόλυτα με τις επιφυλάξεις και τους ε, προβληματισμούς που έχει σημειώσει ο ε, εισηγητής στην έκθεσή του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένα έχει εκφράσει την ανάγκη της δημιουργίας ενός επίσημου νομικού μέσου που θα ρυθμίζει γρήγορα και αποτελεσματικά τη χορήγηση χρηματοοικονομικής συνδρομής στις τρίτες χώρες. Ο κανονισμός όμως άργησε πολύ να έρθει και στο διάστημα αυτό έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα με αποτέλεσμα να μπαίνουν ε, πολλά ερωτηματικά για τη χρησιμότητά του. Και δεν μπορώ να κατανοήσω τη, σκοπιμότητα ενός κανονισμού με τόσο περιορισμένο χρονικό ορίζοντα ε, την ίδια ώρα που και τα επιχειρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν πείθουν ένα άλλο σημαντικό σημείο έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να θυμίσω ότι με τη συνθήκη της Λισαβόνα το Κοινοβούλιο έχει αποκτήσει σημαντικές αρμοδιότητες σε πολλά θέματα και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος στα ζητήματα χρηματοοικονομικής συνδρομής είναι πάγια θέση του Κοινοβουλίου. Έτσι λοιπόν το Κοινοβούλιο θα ήταν δύσκολο να απεμπολίσει αυτό το δικαίωμα ε, οι παρατηρήσεις μου μέχρι τώρα φορούσαν το τεχνικό κομμάτι του κανονισμού. Υπάρχει όμως και ένα ουσιαστικό κομμάτι που έχει να κάνει με την ε, χρηματοπιστωτική κρίση και τη συζήτηση που έχει ανοίξει στο εσωτερικό της Ένωσης για τα θέματα αυτά. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε προς το εξωτερικό σαν τίποτα να μην έχει αλλάξει στην Ένωση. Σαν να μην περνάει η Ένωση μια πάρα πολύ βαθιά κρίση. Δεν ξέρουμε για πόσο θα κρατήσει η κρίση ε, δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε και η αστάθεια των αγορών παγκοσμίω μας καλεί να αντιμετωπίσουμε τα χρηματοοικονομικά ζητήματα συνολικά και όχι με ad hoc αυτό πρέπει να ισχύει εξίσου και για τους εξωτερικούς γείτονές μας που χρειάζονται τη συνδρομή μας. Ο παρόν κανονισμός και αναθεωρήσεις των άλλων χρηματοδοτικών μέσων δεν πρέπει και δεν μπορεί να εξετάζονται σε βραχυπρόθεσμη βάση, αλλά να υιοθετούν μια προσέγγιση για μακροπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη κλίμακα. Τώρα, σε σχέση με τις τροπολογίες που προτείνει ο εισηγητής, συμφωνώ με αρκετές από αυτές, όπως η τροπολογία 2, που διευρύνει το πεδίο εφαρμογής στις χώρες της Κεντρικής Ασίας, την τροπολογία 3 ε, επίσης, που προσδιορίζει ακριβώς το είδος της βοήθειας. Και θεωρώ πολύ σημαντικές τις τροπολογίες 31 και 34 και συμφωνώ πάλι απόλυτα με τον εισηγητή στο θέμα αυτό. Θα ήθελα όμως κάποιες διευκρινήσεις από τον κύριο Καζάκ για τις τροπολογίες 1 και 21 με βάση τις οποίες προσθέτει στον τίτλο ε, τον, ε, στον όρο επιλέξιμες χώρες τον όρο εδάφη. Γιατί μια και στο παράρτημα 1 ορίζονται σαφώς οι χώρες που δικαιούνται αυτής της χρηματοδοτικής συνδρομής και σε αυτό περιλαμβάνεται το κόσοβο βάσει του ψηφίσματος 1244 και τα παλαιστινιακά εδάφη τι νόημα έχει αυτή η τροπολογία και θα ήθελα και τη γνώμη της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με το θέμα αυτό. Τώρα για να τελειώσω, δύο κουβέντες για τη μελέτη που πραγματοποίησε το London School of Economics. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και θα ήθελα να σταθώ σε ένα σημείο, σε ένα συμπέρασμα που έτσι κι αλλιώς και εμείς έχουμε διαπιστώσει στο εσωτερικό της Ένωσης. Όταν υπάρχει οικονομική κρίση, η ταχύτητα αντίδρασης είναι κρίσιμη πρέπει αυτή να αστραπιαία και η εκταμείευση των χρημάτων πρέπει να είναι γρήγορη αλλιώς κάθε βοήθεια χάνει το νόημά της. Αυτά είναι τα σχόλιά μου. Θα επανέλθω με κάποιες ε, τροπολογίες στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. E ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τον εισηγητή και το τμήμα πολιτικής ε, για τη μελέτη που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Γενικό σχόλιο, ξεκινώντας, για το όλο θέμα της οικονομικής αυτής ενισχύσεως. Η χρήση λέξεων εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, καμιά φορά θυμίζει διπλή γλώσσα. Υπάρχουν χώρες και εργαζόμενοι στην Ευρώπη οι οποίοι δέχονται βοήθεια οικονομική και επιβολή άγριων μέτρων λιτότητα και τη μείωση του βιωτικού επίπεδου. Και κατά την άποψή μου, η βάση είναι, προέρχεται απ' έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η λέξη βοήθεια, ενίσχυση, δηλαδή βοηθάει η Ευρωπαϊκή Ένωση άλλε χώρε να αναπτυχθούν. Αλλά κατά την άποψή μου, δεν είναι ελεημοσύνη από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή. Συνδέεται με διάφορε συνθήκε και όρου δεν είναι πολιτικοί όροι της δημοκρατίας αυτοί που επιβάλλονται πολυκομματικών συστημάτων κλπ. που αναφέρονται στα λόγια, αλλά είναι οι όροι δομικών διαθροτικών αλλαγών που επιβάλλει το δούνου του παράλληλα με τις συμφωνίες αυτές υπό την καθοδήγηση της Τρόικας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δείτε το, τη μελέτη στο παράρτημα, κοσυφοπαίδιο στην πρώτη περίπτωση. Όρος 3. Ανάπτυξη στρατηγικών ιδιωτικοποίηση με ενίσχυση τη ε, ε, διακυβέρνηση εταιριών. 6. Επιταχυνθεί η ρευστοποίηση ε, διαφόρων δημοσίων επιχειρήσεων και συνεχιστεί η ιδιωτικοποίηση. Η συμφωνία χρησιμοποιείται σαν ε, όπλο για νεοφιλελευθερισμό και να εφαρμόζεται η οικονομική πολιτική τη δεξιά σε χώρε που χρειάζονται οικονομική βοήθεια. Δεν είναι πραγματική βοήθεια προ αυτέ τι χώρε. Εγώ είμαι αντίθετο προ τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται και λειτουργεί αυτή η βοήθεια όσον αφορά συγκεκριμένα θέματα που αντιμετωπίζουμε. Συμφωνώ με το πνεύμα των σχολείων του κ. Κάζακ. Δηλαδή πρέπει να υπογραμμιστούν τα δημοκρατικά θέματα. Οι όροι αυτοί θα πρέπει να επιβάλλονται πέρα από απλά απλές δομικές οικονομικές πολιτικές. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και αυτές οι πτυχές παραπάνω. Συμφωνώ. Διαδικαστικά μετά. Είμαι υπέρ της μέγιστης δυνατής εποπτείας από πλευράς Κοινοβουλίου. Σημαίνει αυτό συνέχιση της κανονικής νομοθετικής διαδικασίας για κάθε συμφωνία κατά περίπτωση. Τι ο τρόπος θα επιβλέπει ε, καλύτερα την όλη κατάσταση το Κοινοβούλιο. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν το λόγο. Όχι. Άρα μπορούμε τώρα να περάσουμε στο πρώτο σκέλος του σημείου αυτού. Θα ακούσουμε δηλαδή τον καθηγητή Μάικλ Έμερσον. ερευνητής στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικών ε, Μελετών. μας παρουσιάσει λοιπόν την μελέτη του και θα ακολουθήσει γύρω σε ερωταπαντήσεων εφόσον βέβαια οι συνάδελφοι θέλουν να θέσουν ερωτήσεις. Δεν έχουμε βέβαια και πάρα πολύ χρόνο. Παρακαλώ λοιπόν να χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα με τις κονσόλες, οπότε τώρα μπορούμε από την αρχή όμως παρακαλώ να ακούσουμε τον καθηγητή. Θα ξαναβάλω εγώ το χρονόμετρο στο 0. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν κατάλαβα τι συνέβαινε ακριβώς, άρα μου λέτε να ξαναρχίσω από την αρχή. Ωραία. Ναι, υπήρχε ένα πρόβλημα με τις κονσόλες. Παρακαλώ, ξεκινήστε από την αρχή, γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα με τη διερμηνία. Δεν λειτουργήσαν οι κονσόλοι. Α, μάλιστα. Τώρα κατάλαβα, λέει ο κύριος καθηγητής. Φαντάζομαι ότι οι παρόντες ε, γνωρίζουν ε, τι είναι το EPC και τι προσφέρει ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είναι ένας μικρός ε, μέτοχος ε, των ε, πράξεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Κάποιες φορές είναι γύρω στο 10%, άλλοτε λιγότερο. Και αυτό με φέρνει σε ένα από τα πολύ εύστοχα σχόλια της έκθεσης. Νομίζω ότι είναι μία, Τα πάντων, τις τροπολογίες. Πρόσφατα, δύο πράξεις στον χρόνο διεξάγαμε, αλλά όχι με ομαλό τρόπο, διότι αυτό έχει να κάνει βέβαια με τις ε, συνθήκες της οικονομικής κρίσης. Um, <clears throat> on the evaluation of the effectiveness of this instrument, uh, there have been πρόσφατα έγιναν αρκετές μελέτες τις οποίες έχω μελετήσει στη σελίδα 44 της δικής μας έκθεσης. Δεν ξέρω αν έχει διαλλάξει η αρρύθμιση βέβαια. There uh, now it's page, um, έχει αλλάξει η αρρύθμιση. Πρέπει να είναι τώρα 37 38 η σελίδα στη δική σας έκθεση. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι Είδαμε 15 από αυτές τις πράξεις ε, και που καταλήξαμε ότι έξι αξιολογήθηκαν με τον εξής τρόπο. Όχι, εγώ δεν τα λόγω αυτά, κάποιοι άλλοι τα είπαν. Είπαν ότι έχει περιορισμένα μέτρια, μετριοπαθή, λίγα αποτελέσματα, μελιτέα αποτελέσματα. Χρήσιμο που πλευράς απλά προβολής, θα είχε υλοποιηθεί ούτως ή άλλως. Αυτά είναι κάποια από τα σχόλια Άρα μέτρους αντίκτυπος. Δύο πράξεις δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί γιατί υπήρξαν πολύ σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις αλλά υπήρξαν και σοβαρά προβλήματα διακυβέρνησης. Μιλάμε για χώρες όπως είναι η Ουκρανία ή η Βοσνία. Τέσσερις δε εν μέρει ακυρώθηκαν διότι υπήρξε ταχεία μεταβολή των οικονομικών όρων και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην καθίσταται αναγκαία η συγκεκριμένη πράξη, η συγκεκριμένη ενέργεια. Άρα υπήρχαν προβλήματα με την χρονική υστέρηση και την προπαρασκευή των σχεδίων. Κάποια βασικά στοιχεία τώρα, το νέο, ο πλαίσιο που προτείνει η Κομισιόν. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειε γιατί είναι δικό σας ε, καθήκον ε, θεσμικό, θεσμική σας εργασία. Εγώ θα ήθελα να πω ότι η δυσκινησία όλων αυτών των ε, διαδικασιών και οι στερήσεις είναι κάτι που το γνωρίζουμε και κατανοώ ότι πρόκειται για ένα πραγματικό πρόβλημα. Το Σχέδιο κανονισμού πλαισίου προτείνει μεγάλη απλούστευση αυτών των διαδικασιών και από ό,τι γνωρίζω ανθίσταται το Συμβούλιο διατυπώνοντας προτάσεις που τελικά αυτό που σημαίνουν είναι ότι μια Επιτροπή του Συμβουλίου θα επέμενε για την μικροδιαχείριση αυτών των δραστηριοτήτων της Κομισιόν. Άρα ουσιαστικά δεν μπορεί να υπάρξει ταχύτερη διεκπαιρέωση και απλούστευση στις διαδικασίες. Επόμενο σημείο, αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ο μόνος εταίρος για τέτοιες δραστηριότητες, εμείς υποστηρίζουμε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι η κανονική διαδικασία, αλλά όχι η μόνιμη. Δηλαδή, η Παγκοσμία Τράπεζα, η Μπέρντ και άλλοι θα μπορούσαν να συμμετέχουν. Ε, τι είδαμε πριν από κάποια χρόνια στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη με την οικονομική κρίση του 2008 και του 2009. Εθίγησαν πάρα πολλοί χώρες αυτές και τότε κυρίως η Μπέρντ ε, παρενέβη για να βοηθήσει να επιβιώσει το τραπεζικό σύστημα των χωρών αυτών. Και διερωτώ με μήπως με την υφιστάμενη κρίση στην Ευρωζώνη δημιουργηθούν αντίστοιχε συνθήκε και μήπως η Μπέρντ που ξέρει τι ε, κάνει θα μπορούσε ενδεχομένω να παρέμβει και σε αυτή την περίπτωση. Το ερώτημα λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του συγκεκριμένου εργαλείου θα μπορούσε ενδεχομένω να παρεμβαίνει. Και υπάρχουν επιχείρηματα υπέρ αυτής της άποψης. Ένα δεύτερο σημείο που αναφέρει και ο εισηγητής στην έκθεσή του είναι γεωγραφική κάλυψη. Έχουμε τις χώρες της γειτονίας, αλλά γίνεται και μια σαφής αναφορά σε κάποιες άλλες χώρες. Ε, στη δική μου έκθεση, ε, και το λέει και ο εισηγητής να το αναφέρουμε, ε, συγκεκριμένα αναφέρω την Κεντρική Ασία, για να μην είναι σαφής η διατύπωση. Τώρα το θέμα της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και των πολιτικών προϋποθέσεων, political conditionality. Είναι τεχνική ουσιαστικά εδώ η προστιθέμενη αξία, είναι συστήματα ελέγχου των δημοσίων οικονομικών. Ναι, εντάξει, σημαντικό και αυτό, αλλά δεν είναι στρατηγικό. Είναι κάτι που ισχύει σε τεχνικό επίπεδο. Ο εισηγητής λοιπόν προτείνει να έχουμε πολιτικές προποθέσεις, πολιτικούς όρους με πολύ μεγαλύτερη, πολύ πιο ρητά να αναφέρεται. Και αυτό πράγματι συνιστά προστιθέμενη αξία, γιατί το Εθνικό Νομισματικό Ταμείο δεν μπορεί να συμπεριλάβει ρητούς πολιτικούς όρους και προποθέσει, αλλά θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί δεν μπορούμε να αγοράσουμε με 10 εκατομμύρια ευρώ τη δημοκρατία, συνήθω τουλάχιστον. Το θέμα είναι λοιπόν, ή είναι δυνατόν να εντοπίσουμε κάποιες κινήσεις σε πολιτικές ή κάτι, ή θέματα που να έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα. και να ασκήσουμε κάποιε πίεσει, αλλά φυσικά και δεν μπορούμε να αγοράσουμε χονδρικά, αν θέλετε, ε, με κάποια εκατομμύρια ευρώ την ε, βελτίωση πολιτικής κατάστασης και τη δημοκρατία. Ένα άλλο σημείο. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται η εξπόστα αξιολόγηση, δηλαδή εκ των υστέρων αξιολόγηση. Έχω μιλήσει με τον Πίτρε Πέξ από την Κομισιόν και του συναδέλφου του και έχουμε ανταλλάξει απόψει. Η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ε, του συναδέλφου σας αυτού είναι ε, αρμόδια. Έρευνε γίνονται και, από εξωτερικού συμβούλου βέβαια. Αλλά διοντολογικό ε, είναι λίγο αμφισβητήσιμο κατά πόσο ο διευθυντή θα πρέπει να είναι αυτό που αναθέτει τι αξιολογήσει το θέτω απλά υπόψη σε αυτό. Στο Διεθνές Ταμείο και στην Παγκόσμια Τράπεζα οι αξιολογήσεις γίνονται από άλλο τμήμα, όχι από το εκτελεστικό τμήμα ή το τμήμα της διοίκησης. Και ένα άλλο μείζον θέμα, αυτό το μέσο ουσιαστικά μας ε, δείχνει ότι έχει επιτύχει μέτρια αποτελέσματα μέχρι τώρα. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν. Θα πρέπει να πάψει να λειτουργεί, θα πρέπει να επεκταθεί μαζικά η χρήση του ή να το αφήσουμε να λειτουργεί λίγο πολύ όπως μέχρι τώρα. Νομίζω ότι η διακοπή αυτού του μέσου υπό τις παρούσες συνθήκες όταν η Ευρωζώνη πραγματικά ζημιώνει και τους στενούς της γείτονε. θα ήταν κάτι αρνητικό. Θα ήταν πάρα πολύ αρνητικό μήνυμα, πολιτικό μήνυμα άρα δεν είμαστε υπέρ της διακοπής. Τώρα, θα μπορούσε να επεκταθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το μέσο. Γνωρίζουμε ότι η κρίση στην Ευρωζώνη δοκιμάζει ε, τις ε, δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι στα όρια, ίσως έχουν ξεπεράσει τα όρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημείωσα το επιχείρημα του εισηγητή σα ότι η συμβολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η συμμετοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να αυξηθεί κατά τουλάχιστον 20%. το ποσοστό είναι πολύ μικρότερο αυτή τη στιγμή ε, και για το IMF σε σχέση με τον εταίρο αυτό. Άρα ούτε τη δεύτερη εναλλακτική λύση την ε, στηρίζουμε. Δηλαδή ούτε να το διακόψουμε, να το καταργήσουμε, ούτε να το κάνουμε πολύ πιο εκτεταμένο. Αυτό που προτείνουμε είναι να βελτιωθεί αυτό το μέσο, άρα θα βελτιωθεί, πιστεύουμε, και με αυτόν τον κανονισμό πλαίσιο, αλλά και με κάποια από τα άλλα σχόλια που σας ανέφερε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τώρα ερωτήσεις-απαντήσεις. Ας ακούσουμε σχόλια, ερωτήσεις όσον αφορά την παρουσίαση, την ίδια την έκθεση. Μάρτιν, ο εισηγητής μάλλον. Θα μιλήσω βουλγαρικά. Ευχαριστώ. Όσον αφορά το θέμα που συζητάμε, θα ήθελα να πω ότι συγχαίρω καταρχάς τους συντάκτες της ε, μελέτης. Θεωρώ ότι είναι πολύ διεξοδική η δουλειά τους, έξοχη. Τους ευχαριστώ επίσης και την ανάλυση. Είναι πάρα πολύ καλή η ανάλυση του ίδιου του μέσου, του εργαλείου αυτού που γίνεται. Αυτό που προσπαθώ να κάνω, μάλλον προσπάθησα να κάνω, ήταν να εξετάσω με προσοχή τα αποτελέσματα και να τα συμπεριλάβω αυτά τα αποτελέσματα, αυτά τα πορίσματα στη δική μου έκθεση. Αυτές οι συμφωνίες της μικροχρηματοδότησης ήταν κάτι που πάντα συνδεόταν με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όμως, ε, κατά τη δική μου άποψη, όπως και κατά την άποψη διαφόρων ερευνητών, Παραμένει γεγονός ότι πρόκειται περί ενός μέσου το οποίο συνεισφέρει με το δικό του τρόπο. Θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει με το δικό του τρόπο. Δεν μιλάμε μόνο για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα έπρεπε να αναφέρουμε και άλλους εταίρους που υπάρχουν. Όπως είναι η Παγκόσμια Τράπεζα και άλλοι. Ε, στην έκθεσή μου, στο άρθρο 5, 2. πρότεινα μια οριακή τιμή, ένα κατόφλι που σχετίζεται με την βοήθεια που χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε εξαιρετικές ε, περιστάσεις. Είναι ένα όριο το οποίο μπορεί και να μειωθεί. Υπάρχει κάτι που ανέφεραν συντάκτες της μελέτης με το οποίο ε, διαφωνώ. Αυτές οι πολιτικοί όροι, η πολιτική αιρεσιμότητα, αναφέρεται στην επιλεξιμότητα των χωρών η μελέτη. Ε, χωρών που είναι καθοδόν προς εκδημοκρατισμό και προς σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν δούμε ποιοι είναι οι δικοί μας στόχοι, όπως αναφέρονται σε σχέση με τη συνθήκη της Λισαβόνας όσον αφορά συγκεκριμένα τα ανθρώπινα δικαιώματα, αν το δούμε αυτό, τι συμπεριλαμβάνουμε εκεί, πιστεύω ότι βλέπουμε ότι η πολιτική αιρεσιμότητα, οι πολιτικοί όροι που επιβάλλονται στις επιλέξιμες χώρες που είναι αποδέκτες βοηθείας ε, δεν είναι κάτι που συνάδει πλήρως με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δηλαδή, υπογράμμιση, τόνωση των θεμελιωδών αξιών μας. Όσον αφορά τα σχόλια της κυρίας Κοπά, Συμφωνώ με τα περισσότερα που μας είπε και την ευχαριστώ για τα σχόλιά της και ευχαριστώ και τον κύριο Μέρφυ για τις απόψεις που εξέφρασε. Ε, νομίζω ότι κατά τη διάρκεια του διαλόγου μας σχετικά με τις τροπολογίες, κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτών των συζητήσεων για τις τροπολογίες, σίγουρα θα καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία, σε συνένεση. Όσον αφορά το κοσυφοπαίδιο, μια τεχνική διόρθωση έχει γίνει το βρίσκεται διόρθω στο παράρτημα 1. Λοιπόν, όσον αφορά το κοσυφοπέδιο, είναι μία από τις χώρες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, μικροχρηματοδότηση. Όσον αφορά τα σχόλια που έκανε ο κύριος Μέρφυ, όσον αφορά αυτά που μας είπε, λοιπόν, όπου οι ενισχύσεις αυτές θα πρέπει να πηγαίνουν προς χώρες οι οποίες είναι καθοδόν προς μεταρρύθμιση, κυρίως εφαρμόζουν πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Όσον αφορά λοιπόν το θέμα και ότι δεν πρέπει να απειλούμε τις γενικές πολιτικές που εφαρμόζουν αυτές οι χώρες και ότι θα πρέπει να εξυπηρετούμε τους στόχους της κοινωνικής συνοχής και μόνο, αυτός, αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, ένα γρήγορο ερώτημα προς τον καθηγητή. Ποια είναι η άποψή του όσον αφορά την ιδέα διάλυσης του MFA και να ενταχθεί αυτή η ενίσχυση ε, στο μέσο για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία. Να ενταχθεί το μέσο αυτό για τη μικροχρηματοδότηση στην πολιτική γειτονία. Ο καθηγητής ε, κύριος Μάικλ Έμερσον θέλει να απαντήσει στα σχόλια και τις ερωτήσεις που έγιναν. Νομίζω ότι Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή, το MFA, σε κάποιες περιπτώσεις ε, περιλαμβάνει το σκέλος ε, της επιδότησης, της επιχορήγησης, όπως ε, Γεωργία για παράδειγμα η Αρμενία. Νομίζω ότι ο συγκεκριμένο λόγο για του οποίου δίνονται αυτέ οι επιδοτήσει, τα grants, είναι για να ελαφρύνει λίγο του δανειακού όρου σε φτωχέ, υπερχρεωμένε χώρε. Εξού και υπάρχει αυτός ο διεθνής συμπεφωνημένος κανόνας. Αυτό που θα μπορούσαμε να φανταστούμε είναι αυτά τα χρήματα των επιδοτήσεων, των επιχορηγήσεων να μπουν ε, στις επιδοτήσεις ε, της δημοσιονομικής στήριξης που υπάρχει. Θα μπορούσε να γίνει αυτό. Αλλά και από την διασύνδεση με το Διεθνές Ομισματικό Δαμείο. Αν είναι να παραμείνει, ίσως τότε το καλύτερο θα ήταν αυτό να αποτελέσει αντικείμενο ενός ξεχωριστού κανονισμού. Φαντάζομαι όμως ότι και ο κανονισμός ε, για το μέσο γειτονίας, ε, το ΕΝΠΗ, προβλέπει κάποιους μηχανισμούς για τους, με τους οποίους θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά παραπέμπω στην Κομισιόν για το κατά πόσο ε, είναι νόμιμο κάτι τέτοιο ή όχι. Ε, Ολοκληρώσατε, λέει ο Πρόεδρος. Ωραία, σας ευχαριστώ. Ας ακούσουμε λοιπόν τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πίτερ Μπέτσκ. Um, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή σας για την πολύ καλή έκθεση που αποτελεί και μια πολύ καλή βάση για την περαιτέρω συζήτηση. Συμφωνούμε μεν ε, επί σειρά θεμάτων, υπάρχουν ωστόσο και κάποια άλλα θέματα για τα οποία εκφράζουμε κάποιες επιφυλάξεις και ανησυχίες και θα ήθελα τι αρχικέ μου παρατηρήσει να τι εστιάσω σε τέσσερα σημεία. Το πρώτο αφορά τις κατεξουσιοδότηση πράξης. Συμβουλευθήκαμε την νομική μας υπηρεσία για το θέμα αυτό, δηλαδή τη χρήση των κατεξουσιοδότηση πράξεων με την εισαγωγή παραρτήματος, το οποίο θα μπορούσε να τροποποιείται για κάθε απόφαση και η νομική μας υπηρεσία απάντησε ότι είναι ξεκάθαρη η απάντησή τους τέλο πάντων ότι με βάση τη συνθήκη η διαδικασία αυτή τη κατεξουσιοδότηση πράξη εφαρμόζεται μόνο σε μη νομοθετικέ πράξει γενικής εφαρμογή για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση μη βασικών στοιχείων τη νομοθετική πράξη. Αυτά σα τα παραπέμπω όπω τα γράφει ο κανονισμό. Επομένω, να δημιουργηθεί ένα άδειο παράρτημα μόνο και μόνο για να δίνεται στην Κομισιόν δυνατότητα να προσθέτει μια κατεξοδότηση πράξη, τουλάχιστον με βάση την νομική μα υπηρεσία, θα μπορούσε να θεωρεί παράκαμψη τη ε, πραγματική φύση και τη δράση της Κομισιόν, που δεν είναι άλλη από την απλή εφαρμογή του κανονισμού. Ο κύριος ε, Καζάκ αναφέρθηκε ήδη στην γνωμοδότηση της Επιτροπής ΑΦΕΤ και σε αυτό το πλαίσιο το δικό τους επιχείρημα το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Τι λένε λοιπόν, λένε ότι δεδομένου του περιορισμένου εύρους αυτού του μέσου και επειδή πρέπει να είναι αποτελεσματικό και ταχύ, η Επιτροπή ΑΦΕΤ ή τέλο πάντων η εισηγήτρια, κυρία Βάιντερε, στηρίζει την ιδέα να δοθούν εφαρμοστικέ εξουσίε στην Κομισιόν, αλλά προτείνει η διαδικασία των κατεξουσιοδότηση πράξεων να χρησιμοποιείται μόνο στην περίπτωση που θα πρέπει η χρηματοδοτική αυτή συνδρομή να επεκταθεί σε μια χώρα που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των επιλέξιμων χωρών. Και κατά την άποψή μα, είναι ένα αποτελεσματικό τρόπο να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Βέβαια, η Κομισιόν κατανοεί απόλυτα την ανησυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με το δικό του ρόλο θα ήθελα λοιπόν σχετικά να πω ότι οι συνομοθέτες θα διατηρήσουν τον πλήρη έλεγχο του μέσου MFA, της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής. Υπάρχουν όμως και κάποιες εξουσίες προς την ε, Κομισιόν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα μπορεί να ορίζει τους κανόνες και τις προϋποθέσεις για αυτή τη χρηματοδοτική συνδρομή και τον κατάλογο των επιλέξιμων χωρών. Και από εκεί και πέρα, με μονομένες πράξεις, με μονομένες ενέργειες, είναι η, ουσιαστικά η εφαρμογή των κανόνων που έχουν ορίσει από κοινού το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Οι συνομοθέτες φυσικά και θα τηρούνται ενήμεροι για την εφαρμογή τη συνδρομή μέσω των τακτικών εκθέσεων που εκπονούμε για κάθε πράξη, μέσω των ετήσιων εκθέσεων, μέσω των αξιολογήσεων και των λεγόμενων ε, πολιετών ε, αναθεωρήσεων, multi-annual reviews. Υπάρχει διάκριση εξουσιών. Από τη μία έχουμε την εκτελεστική εξουσία, έχουμε την νομοθετική εξουσία και τον έλεγχο από την άλλη. Είναι άλλα τρία θέματα αυτά που θέλω να σχολιάσω, θα είμαι πιο σύντομο για αυτό. Το δεύτερο θέμα αφορά την Κεντρική Ασία ω μια νέα ομάδα επιλέξιμων χωρών. Εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτιμούσε να διατηρηθεί η αναφορά σε άλλε χώρε, other countries. Διότι είναι μεν αλήθεια ότι κατά το παρελθόν η κατηγορία αυτή ουσιαστικά αφορούσε χώρες της Κεντρικής Ασίας, πολύ σωστά το ανέφερε και ο συγητής σας και ο Μάικλ Έμερσον, αλλά τώρα αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη το ίδιο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Την πολιτική δυναμική ε, στις ε, χώρες ε, του Νότου, του Μέσου Γειτονίας. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει ευελιξία για να μπορούμε να βοηθήσουμε τους γείτονές μας, αν υπάρχουν πολιτικοί και οικονομικοί όροι που επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Το τρίτο θέμα είναι το λεγόμενο political conditionality, αυτές οι πολιτικές προϋποθέσεις. Μπορούμε να συμφωνήσουμε με τον εισηγητή ότι είναι καλό να ενισχυθεί ε, αυτό το σκέλος για να έχουμε μια πολύ πιο διαφανή πολιτική αξιολόγηση από την Κομισιόν. Ο εισηγητής προτείνει η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να αξιολογεί την κάθε απόφαση για το κατά πόσον υπάρχει δημοκρατική ευθύνη και λογοδοσία στην εκάστοτε χώρα. Φυσικά, συμφωνούμε και εμεί να συμμετέχει στον έλεγχο των πολιτικών προποθέσεων και όρων και η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Άλλωστε, αυτό πράττουμε ήδη, διότι η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση λαμβάνει μέρο στη διαδικασία λήψεω αποφάσεων που ολοκληρώνεται με την διατύπωση πρόταση από την Κομισιόν διαστόματο υπά τη εκπροσώπου και αντιπροέδρου τη Κομισιόν. Επομένω, επί τη ουσία συμφωνούμε να υπάρχει ένα ρητό, ένα ξεκάθαρο πολιτικό έλεγχο και να ε, πληρούνται κάποιε πολιτικέ προϋποθέσεις. υπάρχει και ένα τέταρτο ζήτημα. Αυτό το θέμα έχει να κάνει το βαθμό στον οποίο η εξωτερική δράση μπορεί να είναι ένα αυτόνομο οργανισμό, μπορεί δηλαδή να ε, αναφέρεται συγκεκριμένα σε μια νομική ε, πράξη. Υπάρχει αυτή η θεσμική συζήτηση η οποία λαμβάνει η χώρα στο πλαίσιο όλων αυτών των συνομιλιών που έχουμε για τα εξωτερικά μέσα του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου. Και εγώ κατανοώ ότι, ίσω βέβαια δεν είναι δική μου αρμοδιότητα αυτό, αλλά εγώ κατανοώ ότι η διασαφήνιση αυτού του νομικού ζητήματο ε, θα επέλθει όπου να είναι, οπότε θα μπορούσαμε ενδεχομένω να υιοθετήσουμε την ίδια λύση που έχουμε υιοθετήσει στα άλλα εξωτερικά μέσα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα δεν είναι αντίθετη με τη γενική αναφορά για πολιτικούς όρους, πολιτικές σε αυτό το μνημόνιο συνεννόησης, αλλά είμαστε κατά του να θεσπιστούν και να καθοριστούν συγκεκριμένα πολιτικά κριτήρια για την εκταμείευση δόσεων της συνδρομής αυτής, γιατί με τον τρόπο αυτό ένα γνήσιο εργαλείο μακροοικονομικής συνδρομής θα μετατραπεί σε ένα πολιτικό εργαλείο, σε ένα πολιτικό μέσο και πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι αντίθετο ε, προς τους στόχους ε, και την αποστολή της ε, χρηματοδοτικής συνδρομής. Το τελευταίο μου στοιχείο έχει να κάνει με την ερεσιμότητα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, IMF Conditionality βοηθά χώρε που έχουν προβλήματα με το ισοζύγιο πληρωμών του στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και δεν μπορεί να το αντικαταστήσει αυτό κάποιο άλλο πολυμερή χρηματοπιστωτικό οργανισμό όπω προτείνεται. Πολύ απλά γιατί δεν υπάρχει άλλο τέτοιο οργανισμό. Δεν παρέχει κάποιο άλλο οργανισμό τέτοιου είδου στήριξη. Όταν ο Μάικλ Έμερσον αναφέρει και στην BERD για τι χώρε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία τη Βιέννη. Ουσιαστικά που είχε ω στόχο να μην αποσυρθούν από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ευρωπαϊκέ τράπεζε. Φυσικά αυτή ήταν μια πολύ χρήσιμη επιχείρηση που είχε πολύ θετικά αποτελέσματα. Αλλά είναι τελείως διαφορετική η φύση αυτή τη επιχείρηση από άλλα ε, δράσεις της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής. Δεν μπορούμε να δεχθούμε λοιπόν, αυτή την πρόταση για τον πολύ απλό λόγο για το ότι εμείς ως Κομισιόν δεν έχουμε πόρους για να αντικαταστήσουμε στα προγράμματα της διαρθρωτικής προσαρμογής, το Διεθνές Ομισματικό Ταμείο. Και άλλωστε εκφίσως από τότε που χρησιμοποιήθηκε, που, που ιδρύθηκε η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή είναι ένα συμπληρωματικό μέσο. Αυτό φαίνεται και από τη διάταξή του και τη δομή του, αλλά και το μέγεθός του. Είναι μικρό μέσο. Ε, δεν ξέρω, θα σταματήσω γιατί φαντάζομαι έχετε και άλλα ζητήματα. αλλά έχω να πω και κάποια σχόλια για πιο τεχνικά θέματα, όχι τόσο σημαντικό σε αυτά τέσσερα που ανέφερα. Ο πρώτος, φαντάζομαι, θα θέλει και ο εισηγητής να σχολιάσει τις ενστάσεις και τα σχόλια της Κομισιόν. Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστώ την Επιτροπή. Αντιλαμβανόμαστε ποια είναι η θέση και η τοποθέτηση της. Με τον κανονισμό αυτό ρυθμίζεται η διαδικασία που αφορά κράτη που μπορούν να επαφεληθούν αυτού του κανονισμού και να εξασφαλίσουν την χρηματοδοτική συνδρομή. Ταυτόχρονα πιστεύουμε και έχουμε και βάσιμα επιχειρήματα, τα οποία άλλωστε έχουμε απευθύνει και στη νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία μας είπε ότι μαζί με τις καταχώρηση πράξεις, το Κοινοβούλιο, με τις καταχώρηση πράξεις, μπορεί, με τις κατεξουδότητες πράξεις, μπορεί το Κοινοβούλιο να συνεχίσει να δραματίσει το ρόλο του, παρακολουθεί δηλαδή και ελέγχει και πόσο σε συνδυασμό με ποιους όρους διατίθενται κονδύλια σε κάποιο κράτος. Αυτή είναι άλλωστε και η εντολή μας. Επίσης, υπολογίζουμε στην υποστήριξη της δανικής προεδρίας για να εξασφαλιστεί μια καλή συμβιβαστική λύση ως έκβαση αυτού του ε, φακέλου της συζήτησης. Καλή λύση που σημαίνει διαφύλαξη της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζουμε ότι θα εξασφαλίσουμε συμβαστική λοιπόν λύση και με, σε συνεργασία με τους κοιόδης συγητές. Σας ευχαριστώ. Καθλώς λέει ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Κλείνει έτσι το θέμα αυτό και η σχετική συζήτηση. 10 Απριλίου, προθεσμία για καταστροπολογιών, το μεσημέρι στις 12 και προτείνω να επιστρέ... επανέλθουμε στο προηγούμενο θέμα. Ναι, και ήρθε τώρα ο εισηγητής. Κύριε Κάσπαρη. Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. με αρμόδια κατ' ουσίαν επιτροπή της, ε, επί της ουσίας επιτροπή, την Επιτροπή Απασχόλησης. Εμείς έχουμε γνωμοδότηση με συντάκτη τον κύριο Winkler, ο οποίος ε, στη συγγνώμη δεν μπόρεσε να έρθει και ζητεί από τον κύριο Κάσπαρη από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να λάβει το λόγο να μας κάνει την παρουσίαση. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να εκφράσω θερμούς χαιρετισμούς από τον κύριο Βίνκλερ, ε, τον συντάκτη, ο οποίος δεν μπορεί να έρθει σήμερα και καθώς το κόλλημα αυτό προέκυψε σχετικά αργά, δεν μπορεί να ε, μεταφερθεί το θέμα στην ημερήσια διάταξη για αύριο. Και μα λέει και ο κύριο Βίνκλερ, λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση συντηρήθηκε το 2007 και εισήχθησαν ε, το 2009 ειδικά μέτρα, τα οποία επεκτάθηκαν το 2011 για να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά προβλήματα της ε, απασχο... που αντιμετώπιζε η απασχόληση στην Ευρώπη. Δε το... Συμπληρώνει μάλλον το Κοινωνικό Ταμείο, το οποίο ασχολείται με τα μακροπρόθεσμα διαρθρωτικά προβλήματα θέματα. Τώρα έρχεται η ώρα της αναθεώρησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Ταμείου αυτού με ε, μία ε, συνθήκη, μία προϋπόθεση για ε, να καταστούν αυτές οι αλλαγές μόνιμες. Θα ήθελα να παρουσιάσω κάποιες από τις προτάσεις μου, από με τις τροπολογίες που έχω προτείνει. Καταρχάς, με το να μείνει έξω από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, εξασφαλίστε μέσω τη προτάσεω. η ε, διαδικασία για κατάθεση των τροπολογιών ε, στο σύνολό της σχεδόν. 11 μήνες δηλαδή θα κρατεί η διαδικασία για να υιοθετηθεί, για να γίνει επεξεργασία μιας αιτήσεως σε παιδοκράτους μέλους. Άρα αυτό μπορεί να οδηγήσει αποτρεπτικά στην αναζήτηση στήριξης από το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίησης Βέβαια θα πρέπει κάθε σημείο της διαδικασίας να επαληθεύεται και να ελέγχεται πολύ προσεκτικά, αλλά θα πρέπει και να υλοποιούνται οι στόχοι του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίησης καθώς ε, δεν αξιοποιούνται επαρκώς κονδύλια υπάρχουν κάποιε επιφυλάξει προ την απορροφητικότητα του Ταμείου και δεν θα ήταν ρεαλιστικό να ζητήσουμε προ χρηματοδότηση και συμπερίληψή του στο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο ήδη από τώρα. Πάντω πιστεύω ότι θα μπορούσαν να περιοριστούν, να περισταλούν οι περίοδοι αναμονή, γιατί περάνε 11 μήνε από την ώρα που καταθέται η αίτηση μέχρι την καταβολή των πληρωμών. Θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει τι διαδικασίε και για την κατάθεση των φακέλων, για την εξέτασή του και για την κατάθεση των ποσών, την διάθεση μάλλον των ποσών. Επίσης φιλοδοξίες και μέσα. Βλέπουμε εδώ κάποια απόκληση καθώς ε, με την πρόθεση της τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να αντιμετωπίσει την απόκληση για περισσότερες επιλέξιμες δράσεις και με μακρύτερη περίοδο χρηματοδότησης. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γεωργοί κυρίως που είχαν de facto αποκλειστεί από την πρόταση του 2007 συμπεριλαμβάνονται πλέον, αλλά ιδιαίτερα οι ε, επιλέξιμοι δικαιούχοι του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα πρέπει ιδιαίτερα να επιλέγονται με βάση το ρόλο που έχει να διδραματίσει το Ταμείο αυτό, δηλαδή προβλήματα κατεπήγοντα, όπως αυτά που θα έπρεπε να υπάγονται στο ε, Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση θα πρέπει να διαφοροποιούνται, να ξεχωρίζουν από τα διαφορετικά προβλήματα ή από, το, ή από τη γεωργία, από τα γεωργικά ζητήματα. Και επίση ε, δεν θα πρέπει αυτό που θα υποφεληθεί από το Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση να υποφελείται από άλλε χρηματοδοτήσει, φερειπίν του Κοινωνικού Ταμείου ή τη ε, Κοινή Γεωργική Πολιτική για του γεωργού. Όλοι οι εργαζόμενοι δε, είτε πρόκειται για εργαζόμενου στην γεωργία, είτε πρόκειται για εργαζόμενου στη βιομηχανία τη υπηρεσία, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ενδέχεται να πληγούν από πολυμερέ ή συμφωνίε, θα μπορούσαν θεωρητικά ανεπάγονται στου δικαιούχου. Εν γέννη, η τάση είναι περισσότερε ρυθμίσει και η πρόταση αναγνωρίζει ρητά πω το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση έχει σαν στόχο την αντιμετώπιση των ε, συνεπειών των Συμφωνίων Ελευθέρου Εμπορίου με μια πολιτική κάπως πιο συσταλτική από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα η Επιτροπή ε, Διεθνούς Εμπορίου θα μπορούσε να δερματίσει πολύ πιο ξεκάθαρα ρόλο στην υπόθεση αυτή γιατί η μέλημά μας είναι και βέβαια οι κοινωνικές συνθήκες ε, εργασίας όσων πλήγονται από την παγκοσμιοποίηση και ιδιαίτερα η Επιτροπή μας αλλά το Κοινοβούλιο και γενικότερα ε, τα ευρωπαϊκά όργανα θα πρέπει να κάνουν μια προσπάθεια να, αντιμετωπίσουν, να βοηθήσουν του ανθρώπου αυτού να αντιμετωπίσουν τι συνέπειε τη παγκοσμιοποίηση. Αυτό είναι και το νόημα των τροπολογιών μου, δηλαδή προσπαθώ να διευκρινίσω του όρου ε, υλοποίηση του Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση και να διευκολύνω τη συμμετοχή σε αυτό των δικαιούχων. Περιμένω να ακούσω τι προτάσει των σκιώδων συγκητών. Αυτά ήταν τα όσα μα ε, προτείνει ο κύριο Βίνκλερ και πολύ ευχαρίστω θα ακούσω τι προτάσει, θα καταγράψω μάλλον τι προτάσει των συναδέλφων μετά τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σαφέστατη η παρουσίαση του εισηγητή. Το σχέδιο εκθέσεως του βρίσκεται στους φακέλους σας με διάφορες ε, τροπολογίες. Πιστεύω κι εγώ ότι η σχέση, ο ρόλος του ταμείου αυτού ε, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της παγκοσμιοποίησης συνδέεται όλο και πιο στενά με την εμπορική πολιτική της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι ασχολείται με τις κοινωνικές συνέπειες εκείνων που πλήγονται από την εμπορική πολιτική της Ένωσης. Η Μαρία Ελένη Κοπά, από τους Σοσιαλιστές έχει το λόγο πρώτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης στην παρούσα χρονική περίοδο είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο δεδομένου ότι μπορεί να στηρίξει τους εργαζόμενους που απολύονται και έτσι να περιορίσει τον αρνητικό αντίκτυπο που έχουν όλες αυτές οι απολύσεις στην τοπική και περιφερειακή οικονομία. Είναι λοιπόν κέρια σημασία η διατήρηση αλλά και η ενίσχυση αυτού του μηχανισμού μέσω της απλοποίησης της χρήσης του και της διάθεσης επαρκών κονδυλίων. Με δεδομένο ότι προβλέπεται η επέκτασή του και στο γεωργικό τομέα που δοκιμάζεται σημαντικά αυτή την περίοδο ε, και λόγω του αντίκτυπου από τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες είναι σημαντικό να παραμείνει ένα έγκυρο και αποτελεσματικό μέσο. Και γι' αυτό η πολιτική μου ομάδα θα είναι υπέρ οποιασδήποτε αλλαγής προς την κατεύθυνση της απλοποίησης της διαδικασίας κινητοποίησης του. Θέλω να τονίσω ότι συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά τη διαδικασία προϋπολογισμού να παραμείνει το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης στα σημερινά δεδομένα. Πρέπει όμως να βρούμε έναν τρόπο οι διαδικασίες να γίνουν λιγότερο χρονοβόρες τέλος θέλω να προσθέσω ότι έχει έρθει η στιγμή να κάνουμε μια σε βάθος συζήτηση όσον αφορά το μοντέλο που χρησιμοποιούμε για τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Πιστεύω ότι δεν έχει καμία αξία να συνάπτουμε εμπορικές συμφωνίες που δημιουργούν ένα μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο και μετά να σπέβδουμε στο Ταμείο Παγκοσμιοποίησης για να περιορίσουμε τις επιπτώσεις. Αυτά είναι τα πρώτα μου σχόλια και επιφυλάσσουμε. Ευχαριστώ. Από τους Πρασίνους, άλλος και ο Ευχαριστώ. Αυτό το ταμείο είναι σημαντικό όσον αφορά την κοινωνική του χρήση. Ακόμα και αν γνωρίζουμε ότι πάνε ένα ταμείο προσαρμογή ε, στην παγκοσμιοποίηση είναι, που χρησιμοποιείται. Κυρίως οι πόροι που χρησιμοποιούνται αντιμετωπίζουν οδηγούνται, ε, δίνονται σε επιχειρήσει που έχουν δυσκολίε όσον αφορά το να λειτουργούν, που δεν σχετίζονται δυσκολίε άμεσα με την παγκοσμιοποίηση. Αλλά υποστηρίζουμε το Ταμείο διότι έχει κοινωνική ε, επίδραση και θέλουμε να προστευτεί η διαδικασία και να επιταχυνθεί. Αντίθετα, εκεί που έχουμε προβλήματα όσον αφορά το θέμα των γεωργών. Ε, βλέπουμε πώς ήρθε αυτή η πρόταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναπροωθεί κατόπιν ιδέας πρωτοβουλία στις διαπραγματεύσεις με τη Μερκοσούρ και βλέπει ότι αυτό δημιουργεί δυσκολίες στα κράτη-μέλη και προφανώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μας δίνει μια πρόταση που είχε σαν στόχο ε, να, να πάει μέχρι τα 2,5 δισεκατομμύρια από τους πόρους αυτούς για να αποζημιωθούν οι γεωργοί που είναι οι πρώτοι που θα πληχθούν από τα αποτελέσματα της συμφωνίας με το Μερκοσούρ. Βλέπουμε ότι γίνονται λιγμοί, κομψή λιγμοί θα έλεγα, αλλά αυτό ήταν ο στόχο, αλλά τελικά τόσο λεπτοί χειρισμοί. Θα γίνουν συμφωνίε ελευθερών συναλλαγών που υπονομεύουν αρκετά σημαντικό τμήμα της Γεωργίας και θα πάμε μετά στους Γεωργού και θα τους πούμε «Κοιτάξτε, ε, κάναμε μια καλή συμφωνία, για εσεί θα εξαφανιστείτε, θα σα δώσουμε μια επιταγή». Ε, και εκτός της ΚΑΠ, εκτός ε, εξέτασης και λήψης υπόψη της γεωργίας στην Ευρώπη. Για μας η ένταξη των γεωργών σε αυτό το ταμείο είναι ένα, αποτελεί ένα διάβημα προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι εντελώς αντίθετη αυτή η πρόταση όχι μόνο έναντι της διαδικασίας μεταρρύθμισης της ΚΑΠ που πρέπει πρώτα να αποφασίσει τι θέλουμε να κάνουμε σαν γεωργία, τι είδους γεωργία θέλουμε, τι είδους γεωργούς θέλουμε να υποστηρίξουμε και εδώ βλέπουμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα διάβημα ε, σχεδόν στρεβλό θα έλεγα ε, ε, θυσιάζοντας τους γεωργούς μας στην Ευρώπη εν ώψη μιας συμφωνίας για ελεύθερες συναλλαγές στον τομέα αυτό με τις χώρες Λατινικής Αμερικής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το πλαίσιο της συζήτησης αυτής είναι ότι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχουμε τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας μετά την εισαγωγή του ευρώ, 25 εκατομμύρια ανέργους. Αυτό είναι αποτέλεσμα της κρίσης, αλλά και η παγκοσμιοποίηση και οι πολιτικές που σχετίζονται με την παγκοσμιοποίηση ευθύνονται γι' αυτό. Άρα στην παρούσα φάση νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε έναν απολογισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση, γιατί έχουμε πολλή εμπειρία συγκεντρώσει. Βάσει των συστήσεων που είχα και με εργαζομένους, οι οποίοι εντός αποφελήθηκαν από αυτό το ταμείο, νομίζω ότι μπορούμε να ότι είναι ανεπαρκέστατο και ακατάλληλο. Και στην πραγματικότητα είναι σαν να βάζουμε χανζαπλάστ ε, σε μια χαίουσα πληγή. Και ίσως γίνει ακόμα χειρότερη κατάσταση με την οικονομική κρίση. Έχουμε τις πολιτικές αυτές ε, που υποτίθεται ότι δημιουργούν απασχόληση, αλλά ε, παρέχουμε ε, κάτι ψίχουλα έτσι μέσω της εκπαίδευσης στον κόσμο, αλλά αυτό δεν ε, αλλάζει την κατάσταση, ότι μειώνω τη θέση εργασίας στην Ευρώπη, ότι υπάρχουν λιγότερες ευκαιρίες για τον κόσμο σε σχέση με τις ευκαιρίες που είχαν παλαιότερα. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένος, υπήρξαν πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν αυτό το ταμείο και δεν είναι ικανοποιημένοι με την εμπειρία. Στην Ιρλανδία υπήρξαν τεράστιες καθυστερήσεις, γραφειοκρατία και η ευθύνη γι' αυτό έγκυται και στην τοπική διοίκηση, στην τοπική κυβέρνηση, αλλά και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ιρλανδία, κατά ε, περίπου το ίμιση των ταμείων που είχαν δοθεί, επεστράφησαν στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν απανήθηκαν εγκαίρω. Όλα αυτά πρέπει να διορθωθούν. Πρέπει να υπάρξει εξορθολογισμό και οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν εύκολα πρόσβαση στα κονδύλια αυτού του ταμείου. Δεύτερον, νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε και λίγο πιο πέρα. Δηλαδή, υπήρξε κάποια παρέκκληση που μείωνε τα κριτήρια της επιλεξιμότητας ε, από τους χίλιους, ανέργου, χίλιους απολυθέντες στους 500 απολυθέντες εργαζομένους και μπλοκαρίστηκε από κάποιες χώρες ε, και από το Συμβούλιο τελικά. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε με το κατόφλι της επιλεξιμότητας και όχι να είναι 500 οι απολυμμένοι, λιγότεροι ακόμη πρέπει να είναι και επίσης το χρονικό περιθώριο, ε, η διορία για την διάρκεια για την οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Ταμείο Εργαζών πρέπει να αυξηθεί. Επίσης πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη συνεκτικότητα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση. Το ένα είναι προληπτικό εργαλείο και το δεύτερο είναι θεραπευτικό εργαλείο, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει συνεκτικότητα ανταγωνιστικότητα μεταξύ τους. Ξέρουμε ότι αυτά τα οποία ισχύουν για το κοινωνικό ταμείο συμμετοχή των συνδικαλιστών κτλ. δεν ε, ισχύουν για το Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Και ένα πολύ επίμαχο κατά την άποψή μου θέμα είναι μείζον συζήτηση που θα γίνει για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και του αγρότε. Ε, κατά πόσο θα μπουν στο Ταμείο ή όχι. Εμεί είμαστε αντίθετοι. Θεωρούμε ότι είναι τελείω χωριστά θέματα. Προβλήματα που δημιουργούνται από την παγκοσμιοποίηση. Χρειαζόμαστε διαφορετικά ε, ταμεία, διαφορετική προσέγγιση. Νομίζω ότι για τους αγρότες καλύτερη λύση είναι μέσω της κοινή γεωργικής πολιτικής να βρεθεί κάποιος τρόπος να αποζημιωθούν. Έχουμε τώρα τις ε, συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών και το λένε πολλοί ότι δεν υπάρχει μέλλον για πολλούς μικρής κλίμακας αγρότες και βάζουμε κάποιους πόρους κατά μέρο για την ε, επανεκπαίδευση, την επιμόρφωσή τους. Όχι, δεν είναι όμως ε, σωστό να ακολουθείτε από την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου αυτή η προσέγγιση. Ευχαριστώ πολύ. Ας ακούσουμε τώρα την Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. προσπαθήσω να δώσω κάποιες απαντήσει για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Το ΕΤΑΦΠΠ δεν αποτελεί αντικείμενο εμπορικών διαπραγματεύσεων. Είναι ένα μέσο, το οποίο στόχο έχει, είναι νομοθέτημα, το οποίο στόχο έχει να βοηθήσει εργαζομένους, τους οποίους έχουν πλήξει διάφορες οικονομικές συνθήκες, και να τους ε, στηρίξει στην ανέβρεση, στην ευχερέστερη ανέβρεση μιας νέας θέσης εργασίας. Στόχο του έχει να εκφράσει με τον τρόπο αυτό την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη εναντί και κάποιων άλλων νομοθετημάτων που το πλήστον είναι εμπορικές συμβάσεις, που, ε, συμφωνίες που ενδεχομένω αποβαίνουν ει όφελο της συντριπτική πλειονότητας των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά που για ορισμένου μπορεί να έχουν αρνητικέ συνέπειε, Εξού και η έννοια τη αλληλεγγύη. Το ταμείο αυτό θεσπίζεται από τα κράτη-μέλη συμπληρωματικά ως προς την εθνική πολιτική που στόχο έχει να βοηθά τους απολυμμένους εργαζομένους. Άρα ε, σέβεται απολύτως την επικουρικότητα στον τομέα αυτό και προσθέτει στοιχεία συμπληρωματικά στις εθνικές δράσεις σε ορισμένες περιπτώσεις. Δηλαδή μπορεί οι εθνικές δράσεις ή να μην υλοποιούνται σωστά ή να μην είναι ορθή η διαχείρισή τους, πράγμα το οποίο μας λυπεί. Πρέπει δεν να σας ενημερώσω ότι η Επιτροπή είχε προτείνει την πρόταση μιας παράτασης ε, κατόπιν των συνεπειών της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης με υψηλότερο ποσοστό, μιας παρέκκλησης μάλλον, με υψηλότερο ποσοστό ε, συμμετοχής, παρέκκληση όμως η οποία λόγω της αντίθεσης ορισμένων κρατών μελών δεν μπορεί να υιοθετηθεί και έτσι δεν ε, ξέφρασαν αντίθεση τα κράτη-μέλη, όπω είπα, και έτσι δεν μπόρεσε να γίνει η διαπραγμάτευση στη συνέχεια με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτήν την έκτατη έκτακτη ρύθμιση, περίοδος 2020 άλλωστε, ε, γνώρισε και αυτή από πλευρά τη την αντίδραση ορισμένων κρατών που την εξέφρασαν την προηγούμενη εβδομάδα με, με επίκληση τη αρχή τη επικουρικότητα, αρχή η οποία είναι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ σημαντική μένα, αλλά από την άλλη ιδιαίτερα θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι του αντίον το ε, δεν παραβιάζει που δεν είναι την αρχή της επικουρικότητας, γιατί κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία υποβάλλουν το σχετικό αίτημα χρηματοδότησης, ε, σε τίποτα δεν τους, δεν τίποτα δεν επιβάλλεται και εκείνα διαθέτουν τα κονδύλια όπως θεωρούν καλύτερο. Μια σειρά τροπολογιών του εισηγητή πρέπει να επισημάνω έχουν ιδιαίτερη αξία και θα πρέπει να τις συζητήσουμε με προσοχή. Εμείς από τις υπηρεσίες επιτροπής του με Ονούς στις προτάσεις του συντάκτη. Επίσης θα ήθελα να πω ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι συμπληρωματικό και ως προς τις εθνικές αρχές, όπως είπαμε, προς εθνικές πολιτικές για την απασχόληση ή την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ενεργείας, αλλά και ως προς το Κοινωνικό Ταμείο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και κατά την υλοποίηση ιδιαίτερα των μέτρων διαπιστώνεται ξεκάθαρα αυτή η συμπληρωματικότητα σε σχέση με άλλα υφιστάμενα χρηματοοικονομικά μέσα. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε αντίθεση, ούτε ασυμβατότητα ή κάποιο άλλο αρνητικό στοιχείο προ την παράλληλη κρίση όπως επισημάνθηκε. Επίσης, θα ήθελα να επισημανώ ότι το να είναι δυνατόν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, ε, προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση, να είναι ανεκτό προς τους ανεξάρτητους επιδευματίες, προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προς τους προσωρινούς, προσωρινώς απασχολουμένους ή απασχολουμένους με ε, σύμβαση ορισμένου χρόνου, επεκτείνει το πεδίο εφαρμογή του Ταμείου σε κάθε τύπο εργαζομένου, πράγμα το οποίο αποτελεί σαφέστατα ένδειξη και αλληλεγγύη, αλλά και ισοδίκη αντιμετώπιση επί Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τελικά σχόλια από πλευρά συζητητού, κ. Κάσπαρη. Ähm, Κύριε Κάσπαρη, Έχω δύο παρατηρήσεις. Ε, υπόθηκε νωρίτερα ότι προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξαναξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις Μερκοσούρ χωρίς να στήσει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μα το Κοινοβούλιο ρητά έχει εκφράσει την υποστήριξή του, κυρία Ζανό, ε, στην επανεκκίνηση, στην ανάληψη των διαπραγματεύσεων αυτών. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα ως προς τις διαπραγματεύσεις. Περιμένω βέβαια να δούμε τι έκβαση θα έχουν και αν θα συζητηθούν τα σημαντικά για εμά θέματα. Αλλά πάντω δεν έχουν κλείσει ακόμα οι διαπραγματεύσει, ούτε και πρόκειται να κλείσουν σήμερα αύριο. Δεύτερον, για τον τομέα τη γεωργία και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη συμπερίληψή του στο Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Ξέρω ότι υπάρχουν ομάδε οι οποίε επισημαίνουν προβλήματα ω προ τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και την συμπερίληψή του εκεί, γιατί γενικότερα ε, τάσσονται περισσότερο προ τι μεγαλύτερε και πιο κεντρικέ δομέ. Πάντω, εμεί πιστεύουμε ότι θα πρέπει οι μικρομεσαίε επιχειρήσει να συμμετέχουν στην παγκοσμιοποίηση. Θα πρέπει να ε, αναγνωρίσουμε ότι ήδη έχουν σημαντική συμμετοχή και φερειπίν παροχή ε, προϊόντων και υπηρεσιών προς μεγαλύτερες ε, παγκοσμιοποιημένες επιχειρήσεις και άρα όταν ε, ε, εκδηλώθηκε η παγκόσμια οικονομική χρηματοπιστωτική κρίση, πολλές από αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάστηκε να απολύσουν υπαλλήλου τους, ανθρώπους που βρέθηκαν στον δρόμο χωρίς κανένα μέσον στήριξης, πράγμα το οποίο δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται δηλαδή ο εργαζόμενος στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει διαφορετική μεταχείριση, γιατί ο ένας ανήκει στην πολυεθνική, έχει απολυθεί από πολυεθνική και ο άλλος έχει απολυθεί από μικρομεσαία επιχείρηση. Αυτό δεν έχει θέση δηλαδή σε μια σύγχρονη και κοινωνική Ευρώπη. Αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω και βεβαίω τι παρατηρήσει των συναδέλφων τι διαβιβάζω στον συντάκτη. Καλώ. χρονοδιάγραμμα. Προθεσμία υποβολή τροπολογιών 29 Μαρτίου στι 6 το απόγευμα. Πάμε στο επόμενο σημείο. Στο σημείο 8 αφορά τον κανονισμό anti-dumping, είναι νομοθετικό θέμα. Είμαστε η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Εγώ είμαι ο εισηγητής. Προσέξτε με σας παρακαλώ. To the Αυτό το θέμα, η άμυνα κατά του dumping, είναι γιατί πρέπει να υφητηθεί σχετικός κανονισμός μετά από την υπόφαση του ΠΟΕ και του Μηχανισμού Διαθέτησης Διαφορών που αποφάσισε ότι όταν διάταξη του κανονισμού δεν συμφωνεί με τους διεθνείς, ότι υπάρχουν διατάξεις που τυχόν δεν συμφωνούν με τους κανόνες του ΠΟΕ. Εμείς υπερηφανευόμεθα που συμμορφωνόμαστε με τους διεθνείς κανόνες εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να ενισχύσουμε την ιδέα κανόνων που εδράζονται επί του συστήματος παγκοσμίου εμπορίου, μας ασκούνται πιέσεις. Μας δόθηκε προθεσμία από το ΠΟΕ μέχρι το φθινόπωρο. Αποφασίσαμε λοιπόν να ακολουθήσουμε τάχιστη διαδικασία. Την απλουστευμένη διαδικασία να ακολουθήσουμε. Άρθρος 46 παράγραφος 1 του εσωτερικού κανονισμού. Αυτό ακολουθούμε. Έγινε διαφωτιστική ανταλλαγή απόψεων με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπάρχει σύμφωνη γνώμη ότι θα πρέπει να θετήσουμε τις αλλαγές που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μας έχουν υποβληθεί. Δεν υπάρχουν πολιτικές διαφορές εδώ. Συμφωνούμε με τους στόχους των αλλαγών όλοι και δεν υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τη διατύπωση της πρότασης. Γι' αυτό προτείνω να ψηφίσουμε ευθύς στην Επιτροπή μας την αλλαγή του κανονισμού άμυνας κατά του ντάμπινγκ Ε, επιταχύνοντας την όλη νομοθετική διαδικασία. Ε, θέλω να ακούσω αν έχετε σχόλια όσον αφορά το θέμα. Η, was... Η απλουστευμένη διαδικασία συμφωνήθηκε, επετέχθη συνένεση στους συντονιστές. Ας ακούσουμε τι έχει να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιος θα μιλήσει εκ μέρους της. Ο κύριος Μάρτιν Λούκας έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προσθέσουμε πολλά στα όσα μας είπατε. Αυτή η πρόταση αλλαγής είναι αποτέλεσμα της προσφυγής της Κίνας στον ΠΟΕ κατά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έχουμε εμεί προσφύγει κατά κινέζικων μέτρων στον ΠΟΕ επανειλημμένα και τώρα εκείνα χρησιμοποιεί το μηχανισμό διαθέσεων διαφορών του ΠΟΕ εναντίον μα. Πέτυχε η προσφυγή τη και πρέπει εμεί τώρα να συμμορφωθούμε με τι υποχρεώσει που έχουμε στα πλαίσια του ΠΟΕ. Δεν κάνουμε τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Χειρουργική τεχνική επέμβαση. Εφαρμόζουμε την απόφαση των δικαστηρίων του ΠΟΕ στη Γενέβη. Αυτά και ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχουν αντιρρήσεις, υπάρχουν επιφυλάξεις, όχι. Οπότε θα κάνουμε αυτό που συμφωνήθηκε. Ψηφοφορία στην Επιτροπή αύριο. Και σημείο 9, πάμε στο σημείο 9, εξωτερική διάσταση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Πρόκειται περί γνωμοδοτήσεως την αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή Αλίας. Συντάκτρια είναι η Ζωζέφα Αντρές. Δεν ασχολείται συχνά η Επιτροπή μας με την αληφτική πολιτική, όμως είναι πολύ εύκολο να καταλάβει κανείς ότι η αλληλευτική και εμπορική πολιτική ε, είναι θέματα αλληλένδετα. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να ασχοληθούμε με το σημαντικότατο αυτό θέμα. Η Ιωζέφα έχει το λόγο, έχει το λόγο Ιωζέφα. Να μας, κάνει μια, να μας κάνεις μια παρουσίαση και να μας παρουσιάσεις την, ε, το σχέδιο γνωμοδότησής σου. Έχετε το σχέδιο γνωμοδότησης του φακέλους σας μονοσέλιδη, μονοσέλιδο κείμενο, έξι παράγραφοι. Έχεις το λόγο, Ιωσέφα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, όπως σωστά είπατε, δεν ασχολούμαστε συχνά με θέματα πάρα πολύ σημαντικά παρόλα αυτά, όπως είναι η κοινή λιευτική πολιτική. Είναι σύντομη η έκθεση, γιατί δεν είχαμε για τις γνωμοδοτήσεις, ε, όπως ήθιστε, παραπάνω χώρο. Προσπάθησα να περιλάβω όμως το θέμα όσο δυνατόν πληρέστερα. Η μετέθεση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και εξωτερική της πτυχή είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους βασικούς ε, πρωταγωνιστές ε, στην διεθνή αλληλευτική σκηνή. Έχει την ευθύνη για την αλληλευτικούς πόρους και την βιώσιμη διαχείριση, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό πρέπει να είναι πυλώνας και της μελλοντικής κοινή αλληλευτικής πολιτικής, όπως και η αρχή της βιωσιμότητας, που θα βασίζεται σε επιστημονικά κριτήρια και θα εφαρμόζονται οι προτάσεις για την ε, πλήρη διαχείριση στο πλαίσιο ενό εργαλείου το οποίο θα καθορίσει ουσιαστικά και το μέλλον ε, τη αλίας. Οι αλληλευτικέ συμφωνίε θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια ρήτρα διαφάνεια στο μέλλον ώστε να μην υπάρχει αλίευση του ίδιου πόρου από περισσότερου ε, του ενό αλληλευτικού στόλους διότι κάποιε φορέ η Ευρωπαϊκή Ένωση με άλλε χώρε ε, που έχουν πιο αρπακτική θα έλεγα διάθεση έρχεται σε αντιπαράθεση. Επίση η αρχή τη Ευθύνη, τη υπευθυνότητα είναι πάρα πολύ σημαντική Πρέπει να ε, καταπολεμηθεί και η άναρχη παράνομη αδήλωτη αλία, ε, IUU όπως λέγεται. Θα πρέπει επίσης να είμαστε ε, ηγετική στην ε, καταπολέμηση αυτή τη αλληλεία και ένα μέρο τη χρηματοδοτική συνδρομή προ τι τρίτε χώρε θα πρέπει να απευθύνεται συγκεκριμένα στην καταπολέμηση αυτή τη μορφή αλληλεία. Γιατί η καταπολέμηση τη παράνομη αυτή αλληλεία θα διατηρήσει βιώσιμε αυτέ τι αλληλευτικέ περιοχέ των τρίτων χωρών. και πιστεύω ότι οι περιφερειακοί οργανισμοί διαχείρισης της αλίας ε, δεν χρησιμοποιούνται ακόμη όσο θα έπρεπε επαρκώς και γι' αυτό θα πρέπει να ε, μείνουμε στο βασικό τους ρόλο και στις εταιρικέ σχέσεις. Οι περιφερειακοί λοιπόν οργανισμοί αλίας θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικά κριτήρια και στοιχεία, σε συνένεση και σωστή εφαρμογή. Οι συμφωνίες είναι μια ασφαλιστική δικλίδα για τη βιωσιμότητα των λευτικών πόρων και είναι πολύ σημαντικό αυτό το κοινοτικό σύστημα ελέγχου του στόλου, βιωσιμότητα και αυτό μπορεί να προσφέρει τα εχέγγυα για τη δραστηριότητα αλλά και τη βιωσιμότητα του αλληλευτικού στόλου. Θα πρέπει επίση να γίνει μια προσπάθεια ώστε οι αλληλευτικέ συμφωνίε με τρίτε χώρε να διατηρηθούν είναι μια εγγύηση για, τη, για το μέλλον της αλίας. Πρέπει, παραλαμβάνω, να καταπολεμηθεί η παράνομη αλία. Εξωτερική διάσταση ουσιαστικά έχει να κάνει με το μέλλον της αλίας και με το μέλλον του αλληλευτικού κλάδου. Θα πρέπει οι αλληλευτικές συμφωνίες να παραμείνουν εγγύηση για τις ε, τρίτες χώρες. Ε, περιμένω και τις ε, τροπολογίες σας για να γίνει ακόμη πιο πλήρης η έκθεση. Με ευχαριστώ. Και τώρα από ο ο Γιάροσλαβ Βαλένσα από το ΕΛΚ. λοιπόν, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Ένα σχόλιο έχω. Νομίζω ότι και στο πλαίσιο του εμπορίου θα πρέπει να προσέξουμε όλος ιδιαίτερος τον αυξημένο ρόλο της επιστήμης στη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί στις διεθνείς προσπάθειες που καταβάλλονται, στους διεθνείς φορείς αλίας, αναφέρθηκαν ε, το, οι διάφορες προσπάθειες που γίνονται. Θα πρέπει να αυξήσουμε, πιστεύω, το ρόλο των περιφερειακών συμβουλευτικών επιτροπών. Θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες, ανεξάρτητες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτως ώστε να ετοιμάζουν ε, ανεξάρτητες γνωμοδοτήσεις. Είναι λόγω επιτροπές έχουν σημαντική τεχνογνωσία όσον αφορά την αλληλεία και νομίζω ότι θα πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την σύναψη νέων συμφωνιών για βιώσιμη αλληλεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Πράσινους, ο Γιάννικ. Ε, δεχόμαστε θετικότατα την παρουσία, στην γνωμοδότηση της συναδέλφου που παρουσιάζει σωστά τα όσα παίζονται στον τομέα της αλληλείας... Ε, και υποστηρίζουμε κυρίως την παράγραφο 6 που έχει σαν στόχο μεγαλύτερη ανιχνευσιμότητα για να σταματήσουν οι εισαγωγές από χώρε που δεν σέβονται τα κριτήρια της βιώσιμης αλίας. Το θέμα της παράνομης αλίας είναι περίπλοκο ζήτημα, διότι η Ευρώπη έχει λίγα μέσα για να μπορέσει στην πράξη να σταματήσει τα ψάρια που προέρχονται από παράνομη αλία. Και αυτό που προτείνουμε ίσως σαν προσθήκη στο κείμενο συναδέλφου είναι να συμπεριλάβουμε την παράγραφο 48 του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Νοεμβρίου του 2011 που λέει ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει συντονισμό και συνεργασία με χώρε που θα μπορούσαν να ε, εφαρμόζουν αυτού του είδου την για να τεθεί τέρμα. Θα μπορούσε επιτέλους να στηριοποιηθεί η Ευρώπη, όχι μόνο στην καταγγελία αυτού του γεγονότος, αλλά και στην πράξη, να εξαφανιστεί αυτού του είδου η αλληλεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Βερόνικα Βάιτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι από την πλευρά μας είναι πολύ ευπρόσδεκτο ότι και αυτή η Επιτροπή ασχολείται με θέματα κοινή αλληλευτικής πολιτικής, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Ένα από τα βασικά στοιχεία που τονίσαμε στην ανακοίνωση για την εξωτερική διάσταση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής ήταν να προσπαθήσουμε να έχουμε μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ κοινή αλληλευτικής πολιτικής και άλλων πολιτικών και κυρίως της εμπορικής πολιτικής Νομίζω ότι είναι σημαντικό να ακούσουμε ποια είναι η άποψή σα όσον αφορά την ανακοίνωση. Τώρα όσον αφορά τη γνωμοδότηση, πράγματι είναι σύντομη, αλλά είναι περιεκτική και όμορφη. Εκτιμούμε τα μάλα τη γνωμοδότηση ως έχει, διότι στηρίζει και πολύ μάλιστα την πρόθεσή μας. Θέλουμε να αυξηθούν οι προσπάθειες όσον αφορά την εξωτερική δράση για, βιο... για βιώσιμη διαχείριση της αλληλείας, σύμφωνα με τις βασικές μας αρχές Δηλαδή, οι όλες οι αποφάσεις για τη διαχείριση της αλληλείας θα πρέπει να σε επιστημονική άποψη και σε παγκόσμιο επίπεδο το ίδιο. Τώρα, αν όπως φαίνεται υπάρξει υποστήριξη της προσέγγισης στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν υποστηριχθεί και η ανακοίνωσή μας, θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Ε, είναι μεγάλος ευρωπαϊκός στόλος, αυτό να το λάβουμε υπόψη και είμαστε από τις σημαντικότερες αγορές για την αλληλεία στον κόσμο. Αν υποστηριχθούμε θα είναι σαφές το πολιτικό μήνυμα. Θα τονωθεί η θέση μας, οι διαπραγματεύσεις μας στο διεθνές προσκήνιο με τρίτες χώρες και θα μπορέσουμε να προωθήσουμε το πρόγραμμα σβησιμότητας και την καταπολέμηση σε παγκόσμιο επίπεδο της παράνομης αλίας. Όπως αναφέρθηκε, υποστηρίζει η γνωμοδότηση τη δημιουργία νέας γενιάς διαφανών συμφωνιών, βιωσίμων συμφωνιών με την αλληλεία, οπότε θα μπορούμε και μακροπρόθεσμα να εξασφαλίσουμε την ε, επάρκεια τροφίμων και να έχουμε και ανταγωνιστικούς αλληλευτικούς στόλους. Τώρα, στην έκτη παράγραφο. Χαίρομαι που η Επιτροπή σας υποστηρίζει την πρότασή μας για εμπορικά μέσα που θα χρησιμοποιούνται σε περίπτωση που δεν αλλιεύουν τρίτα μέρη με βιώσιμο τρόπο. Οι συζητήσει όσον αφορά το εργαλείο, το μέσο αυτό προχωρούν καλά και στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιστεύουμε ότι θα έχουμε ευρία υποστήριξη και από τα δύο θεσμικά όργανα και θα εθετηθεί το μέσο αυτό το ταχύτερο δυνατόν. Και έτσι θα μπορεί να εφαρμοστεί στο εγγύς μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Χωσέφα, μικρή αλλά σοβαρό το περιεχόμενο, μικρή έκθεση αλλά είδατε πόσο την εκθέασε η Κομισιόν, κάτι που δεν συνηθίζει να κάνει. Χωσέφα, συμφωνώ με όλου όσου μίλησαν. Πράγματι, θα πρέπει να φροντίσουμε να είναι εγγύη η Ευρωπαϊκή Ένωση και με τι συμφωνίε που συνάπτει με τι τρίτε χώρε. Θα πρέπει λοιπόν να είναι η πολιτική, όπω είπε και η πρόσωπο τη Κομισιόν, συνεκτική για να μπορέσουμε να συνάπτουμε διαφανεί συμφωνίε, διμερεί συμφωνίε εταιρική σχέση που θα μας δίνουν τη δυνατότητα να βάζουμε όρου προποθέσει, γιατί η αρεσιμότητα είναι και ένα όρο βιωσιμότητα που Μπορούμε να επιβάλλουμε στι τρίτε χώρε. Πιστεύω ότι και η στήριξη τη Κομισιόν αλλά και τα σχόλια γενικά που άκουσα νομίζω θα προσανατολίσουν ε, τη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα κάνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση μεγάλη αλληλευτική δύναμη αλλά και καταναλωτική δύναμη αλληλευτικό Σε ευχαριστώ πολύ, Χωσέφα. Σε ό,τι αφορά τώρα το χρονοδιάγραμμα, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 2 Απριλίου, 12 το μεσημέρι. Έχουμε περιορισμό στο χρόνο μας αφού γνωμοδοτούμε για την ε, καθήλυνα αρμόδια επιτροπή, την Επιτροπή Αλίας και θα πρέπει να βιαστούμε να μην βγούμε εκτός χρονοδιαγράμματος. Ας περάσουμε στο άρθρο στο σημείο 10 και στο σημείο 11 τη διάταξη, τα οποία θα τα συζητήσουμε από κοινού. Η εισηγητή μα είναι ο Χέλμουτ του Σόλτ. Γνωμοδοτούμε για μία επιτροπή, συγκεκριμένα την Επιτροπή Γιούρι και στι δύο περιπτώσει. Η πρώτη έκθεση αφορά την εναρμόνιση Συγκεκριμένα τροποποίηση οδηγία για την αρμόνιση των προθέσεων διαφάνεια αφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότε των οποίων κινητή αξία έχουν την πρώτη διαπραγμάτευση και η δεύτερη έκθεση αφορά τι ρίσκε οικονομικέ καταστάσει, ανοποιημένε οικονομικέ καταστάσει και συναφεί εκθέσει επιχειρήσεων ορισμένων μορφών. Πράγματι σχετίζονται το ένα με το άλλο αυτά τα δύο θέματα, εξού και θα τα συζητήσουμε από κοινού. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας και για τις διεκθέσεις, τον κύριο Χέλμουτ Σόλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, it is really a, quite bigger file. Πραγματικά είναι πολύ ευρύ το θέμα. Η Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου πρέπει να γνωμοδοτήσει για αυτά τα θέματα τα πολύ σημαντικά. Και άλλες επιτροπές γνωμοδοτούν προς την Καθήλυνα Αρμόδια Επιτροπή, την Επιτροπή θα ήθελα να σας παρακαλέσω να συζητήσουμε αυτή τις πολύ στενασυνδεμένες μεταξύ τους προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας περί διαφάνειας έχει ένα γενικό στόχο, δηλαδή να εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνη των επενδυτών, μεγαλύτερη διαπάνεια για θέματα χρεογράφων ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο εισηγητής θέλει να εκφράσει την υποστήριξή του προς μία μείζωνα πτυχή. Δηλαδή, τις απαιτήσει. And logging industry, companies to governments, including in third countries. Και συμπληρωμένο και των τρίτων χωρών σε εξαιρετική βιομηχανία όταν εκδίδουν αξιόγραφα στις διάφορες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, η ετολική σκέψη 14 τη Οδηγία Περιδιαφάνεια του 2004 συνέστησε στα κράτη-μέλη να ενθαρρύνουν τις εισηγμένε εταιρείες των οποίων βασικές δραστηριότητε είναι στην εξορεκτική βιομηχανία να αποκαλύψουν τις πληρωμέ προ κυβερνήσει της ε, τήσιους λογαριασμούς τους και σε εκθέσει τους. Αλλά αυτή η οδηγία επί του παρόντος δεν επιβάλλει υποχρεωτικά αυτό το μέτρο, οπότε τέτοιε πληρωμές που γίνονται σε κυβερνήσει, σε συγκεκριμένε χώρε κανονικά δεν αποκαλύπτουν. Παρόλο που τέτοιε πληρωμέ καταβάλλονται την εξωτερική βιομηχανία. Παραδείγματο χάρη στα ορυχεία, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ε, υλοτομία. Όλα αυτά μπορούν να... Η βιομηχανία αυτή μπορεί να αντιπροσωπεύει σημαντικό τμήμα του εισοδήματο ε, σε χώρε, κυρίω όπω τέτοιε χώρε που είναι πλούσιε φυσικούς πόρους. 3,5 Δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε χώρε των οποίων η οικονομική δομή είναι πλούσια σε φυσικό αέριο, πετρέλαιο και ορυκτά. Η πρόταση για οδηγία για την ετήσια αυτή οικονομική δήλωση, ενοποιημένες δηλώσεις και σχετικές εκθέσεις των διαφόρων επιχειρήσεων. Έχει πολλαπλό σκοπό η προσέγγιση. Πρώτα απ' όλα θέλουμε απλούστευση των διαδικασιών για τις μικρότερες εταιρείες. Δεύτερον, Θέλουμε να αυξήσουμε τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των δηλώσεων αυτών και τρίτον θέλουμε να προστατεύσουμε τις ανάγκες των χρηστών που απαιτούν πληροφορίες ε, λογιστικού τύπου. Τέταρτος στόχος που θα ήθελα να προσέξετε ιδιαίτερα είναι να αυξηθεί η αποκάλυψη, οι απαιτήσει για αποκάλυψη πληρωμών που γίνονται προς κυβερνήσεις από τον εξωτερικό τομέα Παραδείγματο χάρη, επίση και όσου ασχολούνται με την υλοτομία, εταιρείε που ασχολούνται με την υλοτομία. Θέλω να υποστηρίξω αυτή τη βασική πτυχή τη της νομοθετικής Δηλαδή, να υπάρχουν λεπτομερεί απαιτήσει που επιβάλλονται σε αυτές τι εταιρείε, μαζί με την νομοθετική πρόταση περί εναρμονίσεως των απαιτήσεων περί αυτή η νομοθετική πρόταση για τις δηλώσεις οικονομικές θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείε Ευρωπαϊκής Ενώσεως που ανήκουν στον εξορρυκτικό τομέα παρουσιάζουν δημοσία τις πληρωμές προς κυβερνήσεις τρίτων χωρών. Κατά χώρα και κατά πρόγραμμα με λεπτομερή στοιχεία. Επί του παρόντος η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν απαιτεί να αποκαλύπτονται πληρωμές προς κυβερνήσεις που γίνονται σε χώρες όπου εκείνες λειτουργούν. Συνεπώ, αυτέ οι πληρωμέ που γίνονται σε κυβερνήσει συγκεκριμένε χώρε κανονικά δεν ε, κοινοποιούνται. Δημοσίε, πρέπει να δημοσιεύσει αυτά που πληρώνει. Είναι μια αρχή που είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί, ούτω ώστε να επιβληθεί διαφάνεια και να, να ληφθεί η κοινωνική ευθύνη από την εξωτερική βιομηχανία και να μπορούν να ελέγχονται οι κυβερνήσει για τη χρήση των πόρων και να βελτιωθεί η διακυβέρνηση των τρίτων χωρών και έτσι βοηθούμε και την ανάπτυξη αυτών των χωρών. Θέλω οι επενδυτέ τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω να συνεργαστούν στον τομέα τη κοινωνική ευθύνη και να εφαρμόσουν διαφάνεια στη συνεργασία με τέτοιε χώρε. Και πρέπει να δούμε ότι η προμήθεια ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να υπονομεύει τι χώρε που προμηθεύουν την ενέργεια. Η διαφάνεια όσον αφορά τι πληρωμέ προ κυβερνήσει σε αυτέ τι τρίτε χώρε θα συμβάλλει σε καλύτερη διαχείριση των εισοδημάτων που γεννώνται από την εκμετάλλευση των πόρων των αλογοχωρών χάρη σε δημόσιο έλεγχο. Χωρίς έλεγχο δημόσιο, κυβερνήσεις μπορούν εύκολα να ε, μην χρησιμοποιήσουν σωστά αυτούς τους πόρους και να διηγηθούμε σε φτώχεια και συγκρούσεις. Θα πρέπει αυτή η αρχή δημοσίευση αυτά που πληρώνεις να γίνει ένα βασικό εργαλείο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη βελτίωση της διακυβέρνησης. Κάποιοι Επιχειρηματίε θεωρούν ότι αυτό που επηρεάζει σοβαρά την ανταγωνιστικότητα των επενδυτών των Ευρωπαίων στι τρίτε χώρε σε σύγκριση με εταιρείε από άλλε χώρε ε, θα βρεθούν στη δυσχερή θέση διότι έχουν υποχρεώσει περισσότερε και οι άλλοι δεν έχουν ε, τέτοιε υποχρεώσει. Όμω αυτά που διατείνονται δεν υποστηρίζονται δείξει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συμπεριλάβει όμω μια εξαίρεση, ρήτρα εξαίρεση για περιπτώσει συγκεκριμένε, όπου η εθνική νομοθεσία μια τρίτη χώρα κάνει την αποκάλυψη πληρωμών κάτι παράνομο. Ο εισηγητής δεν έχει δυστυχία τέτοιου νόμου που να υπάρχει σε καμιά άλλη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσέξει να μην δημιουργεί ένα κίνητρο για διεφθαρμένες κυβερνήσεις να θεσπίσουν τέτοια νομοθεσία. Επίσης μεγάλες εταιρείες όπως η BP και η Petrobras δεν βλέπουν να υπάρχει ανάγκη μια τέτοια ρήτρα εξαίρεσης. Ας έρθουμε τώρα στις λεπτομέρειες Αντίθετα από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι κανόνες της, ε, των ΙΠΑ που προτείνονται δεν προβλέπουν καμία εξαίρεση πληροφοριών που θα είναι δύσκολο να αποκτηθούν ή να μην αποκαλύπτονται πληροφορίες όταν η, στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα υπάρχει νομοθεσία που απαγορεύει την αποκάλυψη ε, των στοιχείων. Θα πρέπει να αφαιρεθεί αυτή η εξαίρεση από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτω ώστε να ταιριάζουν οι προσεγγίσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των εταίρων μα. Ο ίδιο ο τομέα έχει αναγνωρίσει μέσω τη δική πρωτοβουλία τη διαφάνεια ότι η βελτίωση τη διαφάνεια και του ελέγχου στον τομέα τον εξορυκτικό είναι κάτι που συμβάλλει στην καλή διακυβέρνηση στις χώρες ενεργειακής παραγωγής. Λοιπόν, είναι ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο που θέλει να προωθήσει τη διαφάνεια όσον αφορά το εισόδημα σε κάθε χώρα. 35 χώρες ήδη έχουν ξεκινήσει να εφαρμόσουν αυτή τη συμφωνία, αυτή την προσέγγιση και 60 από τις μεγαλύτερες πετροπολαγωγούς χώρες και χώρες φυσικού αερίου και ε, ορυχείων θέλουν να υποστηρίξουν αυτή την προσέγγιση, αυτή την πρωτοβουλία. Αυτή η πρωτοβουλία έχει υποστηριχθεί πάνω από 80 επενδυτικούς ε, φορείς που συλλογικά διαχειρίζονται πάνω από 16-3 εκατομμύρια ε, δολάρια ήπα. Αρκετές κυβερνήσεις ομάδας των 20, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Διεθνεί οργανισμοί υποστηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε πρόκειται και αυτή να προσχωρήσει αυτή την πρωτοβουλία. Παρόμοια υπόσχεση δόθηκε στη δήλωση της Συνόδου της Ομάδας των 8 στην Τοβίλ τον Μάιο του 2011, όπου οι, ομάδες, οι κυβερνήσεις των ομάδας των 8 δεσμεύτηκαν και παραθέτω να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν νόμους περί διαφανείας και κανόνες σχετικούς για να προωθήσουν εθελοντικές προδιαγραφές που απαιτούν ή ενθαρρύνουν όλες τις εταιρείες εξορρυκτικές να αποκαλύπτουν τις πληρωμές που καταβάλουν προς κυβερνήσεις. Τέλος παραθέσεως. Η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπής, σύμφωνα με το επεξηγηματική της δήλωση, συγκρίνεται ε, με άλλα μέτρα που ελήφθησαν τον Ιούλιο του 2010 στη ΣΥΠΑ και Αφο... Επίσης υπήρχε νόμος του 2010 που θετήθηκε η προστασία των καταναλωτών. και άλλες διατάξεις στον ΙΠΑ προβλέπουν αυτή την προστασία για την εξορυκτική βιομηχανία. Για το πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυκτά. Ορυκτά καύσιμα. Πρέπει να αποκαλύπτουν τα ποσά που καταβάλουν οι κυβερνήσεις. Δυστυχώς δεν έχει ολοκληρωθεί η προσπάθεια στη ΣΥΠΑ. Αλλά υπάρχει δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να ηγηθεί μπορούμε να ενθαρρύνουμε τους βασικούς μας εταίρους στην ομάδα των οκτών να θετήσουν παρόμοια μέτρα. Από τον Ιούνιο του 2010 το Hong Kong επίσης έχει επιβάλει νέους σημαντικούς κανόνες κατά χώρα αναφορά όσον αφορά τις εταιρείε πετρελαίου και ορυκτών καυσίμων που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη έχει περάσει διάφορα ψηφίσματα που δείχνει αποφασιστικότητα όσον αφορά την υποχρεωτική αποκάλυψη πληρωμών που γίνονται στον εξωτερικό τομέα. Τέτοιε απαιτήσει για την αποκάλυψη των πληρωμών συμπληρώνουν την προσπάθεια καταπολέμηση τη διαφθορά μέσω βελτιώσεω των σχέσεων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω με χώρε όπω είναι η Βόρεια Αφρική. Μετά την Αραβική Άνοιξη, την Σαχάρια Αφρική, τη Λατινική Αμερική και αλλού. Εμπόριο, επενδύσεις, όσον αφορά την εξορρυκτική βιομηχανία και θέλω να υποστηρίξω που, ε, ότι ήταν η χαρά μου που ήμουν στην αντιπροσωπεία στις χώρες της Ανατολικής Αφρικής, στην Κένια και στη Ζάμπια πήγα την περασμένη εβδομάδα στις συνομιλίες εκεί. Ε, χαίρομαι γι' αυτό και είναι καλά τα μέτρα αυτά, κυρίως αν λάβει κανείς την οικονομική πραγματικότητα σε αυτές τις χώρες. Εγώ υποστηρίζω ένθερμα τους στόχους της προτάσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όμως είναι καθήκον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου να ελέγξει την πρόταση όσον αφορά την αποδοτικότητα των κανόνων που εφαρμόζεται το διεθνέ εμπόριο. Πρέπει να βασίζεται σε κανόνε και θα πρέπει να θεσπίζουμε νομοθεσίε χωρί να υπάρχουν κενά. Θα πρέπει λοιπόν να διαρωτηθούμε κατά πόσο η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρκετά επακριβής. Παραδείγματο χάρη, είναι αξιέπαινον ότι το σχέδιο οδηγίας απαιτεί κατά χώραν και κατά πρόγραμμα αναφορά. Αλλά ίσως να χρειαστεί να εισαχθεί ακριβέστερη διατύπωση. Τι σημαίνει πρόγραμμα εν τη ενία της οδηγίας. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να αναφέρουμε σαφώς ότι ο όρος πρόγραμμα, project, συμπεριλαμβάνει όλες τις δραστηριότητε που διέπονται από άδεια, εκχώρηση ή συναφή νομική συμφωνία ή αν υπάρχει διαφορετική βάση για ευθύνε, για πληρωμέ, αν υπάρχει διαφορετική βάση και αυτή θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο αναφορά και ενημέρωση. Θα πρέπει να διαρωτηθούμε κατά πόσο το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία είναι παρκέ. Επί του παρόντο, η απόκτηση γεών στον γεωργικό τομέα δεν καλύπτεται. Και αυτό είναι ένα τομέα που δημιουργεί όλο και περισσότερε ανησυχίε. Αλλά επαρκέ. επι του παροντο που κινούνται και δραστηριοποιούνται σε άλλου τομεί όπως λιανεμπόριο, μεταφορές και άλλες δραστηριότητες, ενεργειακή παραγωγή, παραγωγή ενέργειας, που συνεπάγεται αδειοδότηση, ίσως αντιμετωπίσουν αφέμητο ανταγωνισμό από κύριου που μπορούν να καταβάλουν έκτακτε πληρωμέ σε αδειοδοτικέ αρχέ. του ότι τι πληρωμέ είναι ει βάρο των μετόχων. Εάν καλύψουμε κοινοπραξίε επίση, θα πρέπει να τι καλύψουν κοινοπραξίε. Θα ήταν χρήσιμο αν οι εταιρείε θα πρέπει να ανακοινοποιούν τις επιδοτήσεις ούτω ώστε και επενδυτές και η κοινωνία των πολιτών να ξέρουν πού πηγαίνουν τα χρήματα. Θα πρέπει να καλύψουμε τα κενά και θα πρέπει να εξαιρέσει επίσης να εξαλειφθούν. Ο εισηγητής επίσης θα ήθελα να σας καλέσει να επανεξετάσετε τον κατάλογο των απαιτωμένων πληροφοριών προς αποκάλυψη. Ε, οι πληροφορίες αυτές είτε θα χρειαστεί η ΕΣΜΑ ή διάφορες αρχές ελέγχου σε τίτες χώρες ζητούνται πληροφορίες όπως τα κέρδη, όγκοι παραγωγής, εργαζόμενοι, στοιχεία ενεργητικού για να μπορεί να γίνει σωστή αξιολόγηση του εγχειρήματο. Η οδηγία επίση εφαρμόζεται και σε δραστηριότητε εντό Ευρωπαϊκή Ενώσεω και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετίμησε το 2004 ότι η φοραπάτη αντιστοιχεί σε 2,5% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε τέτοια διατύπωση ούτω ώστε να καλύπτουν και την περίπτωση φορολογικών παραδείσων. Θα πρέπει και εκεί που έχουν παρουσία χρηματοστητική εταιρείε να υποχρεούνται να αναφέρουν και πληρωμές σε υποεθνικό επίπεδο και σε δημόσια επιχειρήσει που να καλύπτονται. Και αυτές, αυτά τα στοιχεία τη προτάσεω ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα να γνωστοποιούνται, να ξέρουμε ποια εισοδήματα οι κυβερνήσει αναπτυσσομένων χωρών παίρνουν από τέτοια προγράμματα σε κάποια αιτήματα των χωρών και θα πρέπει να εντοπιστούν περιοχέ οι οποίες δεν ωφελούνται από τα εισοδήματα ε, που παράγονται από τα προγράμματα στη χώρα. Αλλά ποιο ποσό ξεκινά υποχρέωση αναφορά Προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό να εξαρτάται το ποιο ε, καθορίζει το, ε, στην κατ' ουσία νομοθεσία. Οι νομοθέτηση πρέπει να το αποφασίσουν αυτό. Είναι σημαντική πτυχή για να πετύχει η προσπάθεια όλη, το όλο εγχείρημα. Και με αυτά τα εισαγωγικά σχόλια και την ανταλλαγή απόψεων θέλω να σας πω ότι καλείστε τις επόμενες μέρες σε ανταλλαγή απόψεων και συμμετοχή στη θέσπιση αυτής της σημαντικής νομοθεσίας. Προσβλέπω σε επικοδομητική διαδικασία συνεργασίας με τους κοιόδης εισηγητές και θα σας παρουσιάσω σχέδιο γνωμοδότησης 25 Απριλίου, όχι πριν το Πάσχα, αλλά θα είναι προϊόν των πασχαλινών διακοπών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι γνωμοδότηση για την Επιτροπή της. Ας ξεκινήσει λοιπόν η συζήτηση. Έτερος από την Επιτροπή, του συναδέλφους, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, κύριος Αμπάντ. Παρθενική ομιλία στην Επιτροπή μας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Χαίρομαι που είμαι στην Επιτροπή σας για άλλη μια ύστερα από την ε, Επιτροπή των Προπολογισμών, εκπρόσωπο και την κυρία Σάιχη που είναι η συγκεκριτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο και του συναδέλφου από την Σλοβακία που δυστυχώ ούτε ένα τώρα μπορούσε να έρθουν εδώ. Θα ήθελα να πω ότι και οι δύο υποστηρίζουν την πρόταση τροποποίηση τη οδηγία για τη διαφάνεια και την πρόταση οδηγία στη σχετική με, τις, με την υποχρέωση ενημέρωσης των εκδοτών. Δεύτερον, ε, τα θέματα της ε, ενημέρωσης των, ε, του κοινού και ως προς την ενίσχυση βέβαια της κοινωνικής δράσης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και κυρίως αφορά την εκμετάλλευση ορυχείων και δασών σε τρίτα κράτη, σημεία τα οποία ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Επιτροπή μας, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων του 2011 έχει καταγράψει την υποχρέωση για ε, κατάθεση εκθέσεων αναχώρα και ανα πρόγραμμα, οδήγησε σε διάφορα προγράμματα όπως το Flex για τα δάση, για την εξωτερική βιομηχανία όπως επισήμανε και ο εισηγητής. Το άρθρο 6 τροποποιημένο της οδηγίας για την ε, διαφάνεια παραπέμπει ρητά την οδηγία για την ετήσια οικονομική κατασκευή. στο σημείο 9 και γι' αυτό οι σκιώδεις από το ΕΡΚ θα συνεργαστούν στενά. Υπάρχουν διάφορα θέματα προς συζήτηση, διάφορα θέματα που πρέπει να διευκρινιστούν. Φερρυπίν, το πεδίο των δραστηριοτήτων ε, που νοείται εδώ, αν πρόκειται να είναι ημί, οι εκθέσεις της τι είδους πληρωμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν, αν θα πρέπει να προβλεφθεί μια εξαίρεση de ή αν θα πρέπει να δίνονται στοιχεία κατά ε, συγκεκριμένο, άνα συγκεκριμένο έργο. Και αν θα πρέπει να έχουμε ε, διατάξει αντίστοιχες με τις αμερικανικές νομοθεσίες του Frank λαμβάνοντας υπόψη όμως ότι αυτές ακόμη δεν ισχύουν και ότι επιπλέον δεν βρίσκουν ομόφωνη υποστήριξη από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις. Αυτές είναι οι παρέσεις των σχεδόν σύγκητων από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, είναι δικαιολογημένη η απουσία τους και επάξια η εκπροσώπηση τους. Ο κύριος Ντέβιν Μάρτιν, παρακαλώ, στους Σοσιαλιστές Δημοκράτες. Πρόεδρε, ευχαριστώ σκιώδη ηγητή λοιπόν αριστών Δημοκρατών για την οδηγία περί διαφάνεια και θα ήθελα να καλωσορίσω την προσέγγιση του κ. Σόλτ στο θέμα αυτό. Δεν θα ασχοληθώ με τα μη εμπορικά ζητήματα, αλλά μόνο με τα εμπορικά και ιδιαίτερα στην εξωτερική βιομηχανία. Για τα θέματα αυτά λοιπόν θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου για τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κάποιε επιφυλάξει που θα αργότερα. Ε, Πάντω ε, βλέπουμε συχνά ότι η, ο μεγάλος ορυκτός πλούτος των αφρικανικών κρατών αποτελεί πολλές φορές κατάρα και όχι ευλογία, ακριβώς λόγω της εγκατάστασης πολυεθνικών επιχειρήσεων στις χώρες αυτές, οι οποίες πολυεθνικές ε, μεταρχόνται και τα μέσα της διαφθοράς και της πίεσης προς τις τοπικές κυβερνήσεις για να εξασφαλίσουν προνομιακή εκμετάλλευση, ακόμη και βία μεταρχόνται αυτές οι ε, πολυεθνικές επιχειρήσεις και χωρίς βέβαια να ε, αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό απευθείας η σχετική ε, ρύθμιση, πάντως ε, με την εισαγωγή συγκεκριμένων διατάξεων για την χρηματοδότηση μπορεί να επιφέρει περισσότερη διαφάνεια. Η αναφορά, οι καταγραφές δηλαδή εκθέσεων ανά χώρα και ανά έργο είναι πολύ σημαντική. Επεσήμανε ο κύριος Σόλς ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίε. η μία είναι η απόκτηση, δηλαδή όταν μέσα σε μία διαδικασία και ο ζωτικό τμήμα μιας διαδικασίας εξασφαλίζονται συγκεκριμένοι πόροι, γιατί το κύριο και πρώτο βήμα είναι η απόκτηση κυριότητας πάνω στους πόρους αυτούς και καθώς δεν περιλαμβάνεται στη σχετική ρύθμιση ε, βλέπουμε ότι λείπει το κομμάτι αυτό. Επίση, η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. Πολλέ είναι πολυεθνικέ οι οποίε έχουν προσυπογράψει θετικέ ε, ρυθμίσει, χωρί όμω ε, να τηρούν, όπω διαπιστώνεται εκ των υστέρων, τι υποχρεώσει του και πώ ξεφεύγουν από αυτήν την υποχρέωση, αναθέτοντα σε υπεργολάβου την εκτέλεση του έργου. Άρα, θα πρέπει όχι μόνο η πολυεθνική απευθεία, αλλά και το τρίτο μέρος το οποίο αναλαμβάνει εξ ονόματος τη Πολυεθνική να εκτελέσει έργο, να υπολογίζεται σε αυτή την τήρηση της κοινωνικής, των όρων τη κοινωνική ευθύνη. Δεν θα είπε αυτέ τι λεπτομέρειε γιατί δεν έχουμε χρόνο, αλλά πάντω είναι πολύ καλέ εξελίξει, θετικέ εξελίξει και περιμένουμε να δω και το γραπτό κείμενο για πιο συγκεκριμένε προτάσει που θα οδηγούσουν προ την υλοποίηση του. Ευχαριστώ. I have no more for the Θέλει κάνει άλλο το λόγο, παρακαλώ. Ας ακούσουμε και την Επιτροπή αν είναι έτοιμη. Υπάρχει εκπρόσωπος της Επιτροπής για κάθε ένα από τα κεφάλαια, τη διαφάνεια, οδηγία για τη διαφάνεια. Κύριε Αντικολομπιέ. Ε, actually, the... Feel free. Yes. Ε, Όχι, ελεύθερα, ελεύθερα αρκεί να μας πείτε, να μας πείτε ότι εκπροσωπείτε την Επιτροπή. Μάλιστα κύριε Πρόεδρε, ε, και για, τους, για τις δύο οδηγίες έχουμε εκπροσώπους εδώ. Εγώ όμως θα να αναφερθώ κυρίως στην έκθεση χώρα» και μια και τα περισσότερα σχόλια αφορούσαν το κομμάτι αυτό. Θα ήθελα να απαντήσω. Καταρχάς ευχαριστώ όλους τους ομιλήσαντες για, τις, ε, για τα σχόλια. Ο εισηγητής κύριος Σόλτς νωρίτερα επεσήμανε την παρέκκληση που έχει εισαγάγει στην πρόταση της Επιτροπή. Παρέκκληση βάσει τη οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει πολύ περιορισμένη παρέκκληση για να προστατεύει εργαζομένους ε, που εργάζονται ε, επιχειρήσεις ε, από την, τους απαλλάσσει από την υποχρέωση αποκάλυψης εσόδων ή μάλλον αμοιβών, ώστε να μην εκτεθούν σε ποινική ε, δίωξη λόγω αυτής της αποκάλυψης στοιχείων. Δεν θέλω να σας ενημερώσω, είναι μια πολύ περιορισμένη παρέκκληση. Θέλουμε να προστατεύουμε τους ε, απασχολουμένους εφόσον υπάρχει πρόβλημα με την νομοθεσία της χώρας. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε συναντήσει όμως. Πάντως, ε, εάν την παρέκκληση αυτή την επικαλεστεί κάποια πολυεθνική, θα πρέπει να λέει και σε ποια χώρα αναφέρεται η παρέκκληση. Για τον νόμο Dot Frank που ε, επεσήμαναν αρκετοί βουλευτέ. Οι προτινόμενε διατάξει ακόμη δεν έχουν ακόμη τελειοποιηθεί. Αναμένονται τον Ιούνιο του 2012 και ω εκ τούτου δεν γνωρίζω ε, εάν και εφόσον θα προβλέπουν παρακλήσεις στον τομέα αυτό. Πάντως, έχουμε μια γενική εικόνα για τον νόμο Dodd Frank, αλλά δεν ξέρουμε αν στους, ε, εάν θα επισέλθει σε αυτή τη λεπτομέρεια προς τους εφαρμοστικούς κανόνες. Επίσης, συμφωνώ με τον εισηγητή ε, στην παρατήρηση ότι θα πρέπει οι χωρε g G8 να ενθαρρυνθούν για υψηλότερες, με προσπάθεια για υψηλότερες Πρόκειται για προδιαγραφέ σημαντικέ όχι μόνο για τι αναπτυσσόμενε χώρε. Αλλά θα ήταν αυτό ένα βήμα σημαντικό και για την ανταγωνιστικότητά μα, γιατί η αποκάλυψη πληροφοριών θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκάλυψη και ευαίσθητων πληροφοριών. Άρα θα πρέπει όλε οι χώρε, όλε οι επιχειρήσει μάλλον να υπάγονται ε, στους ίδιους κανόνες και εμείς θα ενθύρναμε μάλιστα τις ε, χώρες του G20 να ενθαρρύνουν τις, ε, να, να ακολουθήσουν τις προδιαγραφές αυτές. Για τον προσδορισμό των έργων, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι έργο ως όρος συνεπάγεται τρεις διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας. Την εξορρυκτική που περιλαμβάνει και τα ορυχεία βέβαια αλλά και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, την ε, δασοκομεία και έτσι προσπαθούμε να βρούμε από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ορισμούς ικανούς να καλύψουν κάθε τύπο δραστηριότητας γιατί βέβαια ε, εξωτερική βιομηχανία, εξωτερικό κλάδος καλύτερα μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε κάθε χώρα. Φερρυπίν, μία επιχείρηση μας είχε πει ότι ο όρος ε, έργο στον Καναδά μπορεί να σημαίνει πολύ μικρά μόνο τεμάχια. Ενώ η χώρα αυτή, ενώ η επιχείρηση αυτή μάλλον, είχε 10.000 τουλάχιστον εκμισθώσεις στον Καναδά, ενώ σε μια άλλη χώρα είχαν μόνο δύο εκμισθώσεις γης η εκμετάλλευση. Εν πάση περιπτώσει, εάν ακολουθήσουμε τη μέθοδο αυτή, θα πρέπει να ε, καταλήξουμε σε φερειπίν στη συγκεκριμένη περίπτωση 2.000 διαφορετικές εκθέσεις ε, το, με, με, συνέπεια μεγάλο γραφειοκρατικό φόρτο για την επιχείρηση. Άρα θα πρέπει να βρεθεί μια λύση λογική που θα επιτρέπει στην ε, επιχείρηση, στην λόγω επιχείρηση να ακολουθεί το εσωτερικό της σύστημα καταγραφής εκθέσεως στο χαμηλότερο του επίπεδο. Ακολουθεί τη δική της δομή δηλαδή. Για τους τομείς θα μπορούσαμε να έχουμε προχωρήσει περισσότερο. Βέβαια, στόχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν περισσότερο να στηρίξει, να ενισχύσει περισσότερο οι υφιστάμενες ε, διεθνείς πρωτοβουλίες Όπω η ITI που αφορά κυρίως τον εξωτερικό κλάδο, και ξέρουμε ότι στη Λιβερία Φερρυπίν γίνεται αποκάλυψη στοιχείων και για τον χώρο της νοσοκομεία. Επικεντρωνόμαστε σε αυτού του τομείς γιατί πρόκειται για μία ανανεώσιμε πηγές που ανήκουν στο λαό και που έχουν μεγάλη σημασία για τι αναπτυσσόμενε χώρε. Τι γνωρίζουμε σε ορισμένε χώρε ο εξωτερικό κλάδος ε, εξασφαλίζει έως και 50% των εσόδων του γενικού κράτους και πολύ μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ σε ορισμένε αφρικανικές χώρες. Η Επιτροπή έχει εισαγάγει στην πρόταση και ρήτρα που θα επιτρέπει την δυνατότητα σε μια παρέξεταση να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής αφού αναθεωρηθεί η λειτουργία της προτάσεως. Επίσης, τελευταίο στοιχείο, το σχετικό με τις ε, κατεξουσιώτες πράξεις και τον ορισμό των ορίων, των κατοφλίων δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι δεν ήταν ευχαίρες ε, το να προσοριστεί ένα κατόφλι υλοποίησης και έτσι προτείναμε τη λύση, για να κερδίσουμε χρόνο, τη λύση της κατεξουδότησης σύμπραξης. Αυτό ήταν το νόημα μόνο. Ευχαριστώ. Καλώς, λίγο Πρόεδρος. Άλλες παρατηρήσεις. Όχι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ναι, και για τη διαφάνεια και για τις ε, εκθέσεις ήταν αυτό, Πρόεδρε. Μάλιστα, επομένως, μπορούμε να συνεχίσουμε πανερχόμενοι στον εισηγητή, e e κύριο Σόλτς. Uh, thank uh, Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άκουσα τους συναδέλφους, άκουσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθώ τη δουλειά αυτή και, στους, και στους δύο τομείς. Θα επανέλθω μάλλον στη συζήτηση και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα άρθρα 38 και ιδιαίτερα στην παράγραφο 5 όπου θα μπορέσουμε να δούμε αν βρίσκεται λύση που να καλύπτει και τις λύσεις του David Μάρτιν από τους σοσιαλιστές δημοκράτες και τις παρατηρήσεις του. Θα ήθελα επίσης να πω ότι είναι σημαντικά αυτά τα θέματα. Θα προσπαθήσω, όπως είπα, να συντάξω το σχέδιο. Mr. Lehne concerning the whole um, um, issue And so we have to see what is the opinion also of the other committees and so that the time frame which is foreseen for adopting of the dossier. Και το χρονοδιάγραμμα που χρειάζεται να τηρηθεί. Ιούλιο, Σεπτέμβριο στην Ολομέλεια. Καλώς, ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. 10 Μαΐου, 6 το βράδυ, προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών. Εδώ τελειώνει το δημόσιο τμήμα της συνεδριάσεως μας σήμερα. Θα συνεχίσουμε με συντονιστές και ως εκ τούτου παρακαλώ ή ονδήποτε δεν έχει σχέση με την συνεδρία των συντονιστών να αποχωρήσει το ταχύτερο δυνατό από την αίθουσα.